Bonjour. Eh bien... Χαίρετε και καλώς ήρθατε όλοι. Αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις ή σχόλια όσον αφορά το σχέδιο ημερησίας διατάξεως. Παρακαλώ, εάν όχι, εγκρίνεται λάβατε και τα πρακτικά της συνεδρίας της, της 5ης Νοεμβρίου 2012. Αν έχετε παρατηρήσει σχετικά με τα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής, παρακαλώ να ενημερώσετε τη γραμματεία μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αυτή. Διαφορετικά τα πρακτικά αυτά θα εγκριθούν. Έχετε λάβει στους φακέλους σας τις συστάσεις και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση των συντονιστών στις 21 και 10... Ε, Νοεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου. Αν έχετε σχόλια σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της συνεδρίασης, παρακαλώ να το επισημάνετε πριν από το πέρας της συνεδρίασης αυτής. Εάν όχι, τα αποτελέσματα αυτά θα υιοθετηθούν ως έχουν. Εγώ δεν έχω άλλα σχόλια ή ανακοινώσεις να σας κάνω. Η Επιτροπή έχει κάποια ανακοίνωση να μας κάνει. Όχι. Δεν έχουμε λάβει ερωτήσεις που θα πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω την ευχαρίστηση να υποδεχθώ τον Επίτροπο Κίμπαλξ για μια πρώτη συζήτηση στο πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης. Θα ανταλλάξουμε απόψεις επί του προγράμματος εργασίας του 2013 ε, όσον αφορά την πολιτική της ανάπτυξης. Ε, πρόκειται για αυτό που αποκαλούμε διαρθρωτικό διάλογο. Κατά τον ίδιο τρόπο, αύριο θα έχουμε έναν διαρθρωτικό διάλογο με τον Επίτροπο Ζόρσεμπα όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Επίτροπε και σας δίνω αμέσως το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ε, προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω ένα, ε, μια σύνοψη της πρόοδου που σημειώσαμε ε, φέτος και να εξετάσω μαζί σας τις προοπτικές για το προσεχές έτος. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι το 2012 ήταν ένα μάλλον καλό έτος για την πολιτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις τεράστιες προκλήσεις, μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε ευρεία αποδοχή για την ατζέντα της αλλαγής και την ε, νέα ανεπτυξιακή πολιτική. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να ε, μπορέσαμε να χορηγήσουμε βοήθεια με πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Αυτά είναι ευχάριστα νέα. Η ατζέντα λοιπόν για την αλλαγή του Συμβουλίου συνδυάστηκε με το γεγονός ότι και πολλές χώρες μέλη έχουν μια παρόμοια προσέγγιση στο θέμα της συνεργασίας. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση διατήρησε τον ρόλο του ηγέτη στις διεθνείς εξελίξεις σε αυτό το, έ το Διεθνές Έτος Βιώσιμης Ενέργειας για Όλους έχει αναγνωριστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε έναν κυρίαρχο ρόλο ως προς την ατζέντα αυτή. Τούτο συνέβαλε στο να δημιουργηθεί μια διεθνή συμμαχία βασισμένη σε εταιρικέ σχέσεις ε, και έτσι δημιουργήθηκε ένα δίκτυο επένδυσης υπέρ του κλίματος αλλά και χωρών δωρητών ώστε να χρηματοδοτηθεί αυτό το καινοτόμο χρηματοδοτικό μέσο που θα χρηματοδοτήσει τις ε, σύγχρονες πηγές ενέργειας έως το 2030. Η διάσκεψη, στη διάσκεψη κορυφής τον Απρίλιο, ο πρόεδρος Μπαρόζο είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει 500 εκατομμύρια ανθρώπους να εξασφαλίσουν βιώσιμη ενέργεια μέχρι το 2030. Κανένας ε, δεν Ισχυρίζεται ότι αυτό είναι κάτι απλό. Αντιθέτως, πρόκειται για τεράστια πρόκληση. Ωστόσο, είναι μια πρόκληση που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση ε, να αντιμετωπίσει. Η αποφασιστικότητά μας ε, να υποστηρίξουμε τη βιώσιμη ενέργεια για όλους ε, αντανακλάται σε όλα όσα κάνουμε μέχρι στιγμής με τον ίδιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να προχωρήσει και στο θέμα της διατροφής. Ε, διαδραματίζουμε λοιπόν ηγετικό ρόλο και στο θέμα αυτό που βασίζεται σε παρόμοιες αρχές με αυτές της βιώσιμη ενέργειας και ήδη αποδίδει παρόμοια αποτελέσματα. Ε, βέβαια, ως προς τα επίπεδα βοήθειας που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητικά. Για πολύ κατανοητούς λόγους, ε, πολλές χώρες έχουν μειώσει τις φιλοδοξίες τους. Έχουμε λοιπόν 0,7% αυτού που υποσχεθήκαμε. Και ε, ελπίζουμε ότι οι χώρες μέλη θα μπορέσουν να διαθέσουν το δικό τους μερίδιο με βάση το εισόδημα από τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ωστόσο, ισχυρίζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρήσει αυτή τη δέσμευση, όπως ακριβώς δεσμεύθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φέτος. Αν λοιπόν το 2012 ήταν ένα καλό έτος, Έχω τη φιλοδοξία το 2013 να είναι ένα έτος καμπή, διότι η ατζέντα για την αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή. Δηλαδή, θέτουμε το στόχο για την βιώσιμη ανάπτυξη προς όλους, για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Η ε, βοήθεια, η αρρωγή μας θα είναι ο καταλήτης για την αλλαγή της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Βοήθεια, αρρωγή με σημαντικές συνέπειες και που θα στοχεύει αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο και θα είναι όσο πιο αποτελεσματική γίνεται, ώστε να έχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα εκεί επί τόπου και να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα χρήματα που ξοδεύουμε. Έτσι λοιπόν απαιτείται συνεργασία και από κοινού ε, προγράμματα με τις χώρες ετέλους. Παράλληλα με την ατζέντα για την αλλαγή, η εξυγχρονισμένη προσέγγιση μας για την εφαρμογή του προϋπολογισμού αποτελεί ε, κυρίαρχο στοιχείο ώστε οι πολιτικές μας να αποδίδουν καλύτερα μειώσαμε την υποστήριξη, την οικονομική στήριξη προς τις ε, χώρες μέλη. Από την άλλη απαιτείται υψηλού επίπεδου διακυβέρνηση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα έχουμε επιπρόσθετη υποστήριξη του προϋπολογισμού ώστε να επιτευχθούν μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς και να υπάρχουν πραγματικά αποτελέσματα. Επίσης θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις χώρες που βρίσκονται σε εύθραυστη κατάσταση ή σε μεταβατική φάση. Υπάρχει μια νέα μορφή ε, βοήθειας που βοηθά ακριβώς τους ζωτικούς τομείς αυτών των κρατών. Έτσι λοιπόν, η υλοποίηση αυτών των βασικών αρχών, το τα προσεχή χρόνια θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση, να έχουμε μια πιο προβλέψιμη και πιο αποτελεσματική δημοσιονομική υποστήριξη. Ε, πέρσι, τέτοια εποχή, σας παρουσίασα τις προτάσεις της Κομισιόν για την εξωτερική ε, βοήθεια. Θα σας απογοήτευα αν η πρότασή μας για μια σημαντική αύξηση του DCI και του EDF δεν εξασφάλιζε την αποδοχή, την απαιτούμενη αποδοχή. Έτσι λοιπόν κάνω έκκληση να κρατηθούν όλα αυτά τα επίπεδα, ε, όλα αυτά στο επίπεδο που επιθυμούμε. Και γι' αυτό βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη για να με βοηθήσετε να πετύχω αυτό το σκοπό. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω στο λεπτό θέμα των ε, δράσεων που ανατίθενται σε τρίτους. Ε, βασικό θέμα είναι ο δημοκρατικός έλεγχος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες αφενός και ένα ευέλικτο λειτουργικό σύστημα αφετέρου. Πιστεύω ότι αυτό θα αποδώσει. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεργαστώ μαζί σα και με του συναδέλφου του Συμβουλίου τη Προσεχή Εβδομάδα ώστε να βρούμε τη σωστή ισορροπία ω προ την εμπλοκή του Κοινοβουλίου στο πρόγραμμα αυτό. Επιτρέψτε με τώρα να έρθω σε ένα άλλο θέμα ε, δηλαδή το πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015. Η Κομισιόν εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία περιγράφει ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χαράξει την πολιτική της με βάση τους στόχους της μετά το 2015 και τους στόχους ανάπτυξης δηλαδή της χιλιετίας. Ε, στη συνεδρίαση της, ε, του Σεπτεμβρίου ε, ένα, θα υπάρξει συγγνώμη, μια ευρεία έκθεση σχετικά με το τι επιτύχαμε ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Και επίσης θα υπάρξει μια έκθεση από την ομάδα ε, που ασχολήθηκε με την ομάδα εργασίας που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και στις αρχές του προσεχούς έτους θα σας στείλω λεπτομερό στο περιεχόμενο της έκθεσης αυτής αλλά θέλω να σας δώσω κάποιες ε, γενικές αρχές. Βασική μας προτεραιότητα θα πρέπει να είναι μια νέα όθηση στα προγράμματα ε, για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Ιδιαίτερα προς τις χώρες εκείνες που το έχουν ανάγκη. Οι αναπτυξιακοί στόχοι χιλιετίας MDGs λοιπόν νομίζω ότι στέφθηκαν με επιτυχία και γι' αυτό δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να σταματήσουν. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε ότι ο αγώνας ή μάλλον ο πόλεμος κατά της φτώχειας ε, δεν έχει φτάσει στο τέλος του. Αντιθέτως, πρέπει λοιπόν να δράξουμε την ιστορική ευκαιρία που έχουμε στα χέρια μας, ώστε να εξαλείψουμε τη φτώχεια κατά τη διάρκεια της δικής μας γενιάς. Δεν θα είναι κάτι εύκολο. Απαιτείται όμως αποφασιστικότητα για να το επιτύχουμε. Άρα λοιπόν η αφοσίωσή μας σε αυτό θα πρέπει να είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Η εγγύηση μιας αξιοπρεπούς ζωής για όλους μέχρι το 2020 θα πρέπει να είναι το όραμά μας. Η μετατροπή του στην πραγματικότητα απαιτεί να επιλύσουμε θέματα ανθρώπινης ανάπτυξης και άλλων βασικών θεμάτων. Θα πρέπει να επιδιώξουμε ώστε και οι κρατικοί φορείς και οι διεθνείς φορείς να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο για όλους τους πολίτες πάνω στο πλανήτη. Τα αποτελέσματα θα πρέπει οι πολίτες όλου του κόσμου να τα απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις τους και τους ηγέτες τους το αργότερο μέχρι το 2030. Επιπλέον, οι εύθραυστες και ευάλωτες χώρες θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερα επίπεδα ζωής και να ξεπεράσουν την ανασφάλεια και τη βία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η δεύτερη αρχή θα πρέπει να είναι η εγγύηση της δημοκρατίας αλλά και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανάπτυξη της ευημερίας και η ανάπτυξη νέων θέσεων απασχόλησης. Δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπή ζωή από μόνο της. Η τρίτη αρχή που θέλω να τονίσω είναι η καλή διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως επίσης και το εισόδημα από τους φυσικούς πόρους, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του περιβάλλοντος και να υπάρξει μια ισότιμη μεταχείριση και χρησιμοποίηση. Είναι καιρός να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον με βιώσιμες πρακτικές πριν αυτές απειλήσουν το μέλλον, ε, το μέλλον μας. Αυτές οι βασικές αρχές βρίσκονται κάτω από τις φιλοδοξίες που έχω. Με βάση αυτό λοιπόν ε, τρεις διαστάσεις βιώσιμης ανάπτυξης που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ατζέντα μετά το 2015. Παρόλο που δεν εξασφαλίζεται η απόλυτη επιτυχία, πάντως Υπάρχει μια σημαντική πρόοδος. Η παγκόσμια ε, αηφορία και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι βασικά στοιχεία, ενώ η καταπολέμηση της φτώχειας ε, είναι το τρίτο στοιχείο. Η κλιματική αλλαγή, μια άλλη βασική πρόκληση, θα ε, πλήξει τις περιοχές εκείνες που είναι οι περισσότερο ευάλωτες. Και εμείς όπως και η διεθνή κοινότητα συμφωνήσαμε ότι οι βιώσιμοι στόχοι θα πρέπει να είναι συνεκτικοί και να συνδυάζονται και με την ολοκληρωμένη ατζέντα μετά το 2015. Αυτή η διαδικασία λοιπόν θα πρέπει να γίνει με συντονισμένο τρόπο ώστε να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να διαδραματίσει έναν κυρίαρχο ρόλο και πιστεύουμε ότι οι δύο αυτοί παράλληλες οδοί θα πρέπει να προχωρήσουν ε, παράλληλα. Θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή αυτή και η συμβολή της θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Επίσης, θα εστιάσουμε την προσοχή μας και σε σειρά ε, εκδηλώσεων που θα οργανώσουμε του χρόνου για να εμπλέξουμε και την κοινή γνώμη. Άρα, τα βασικά παραδοτέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική ανάπτυξη μέχρι το 2030 θα είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζουν την υλοποίηση της ατζέντα και να διασφαλίζουν ότι η φωνή της Ευρώπης θα είναι ισχυρή και ενιαία σχετικά με την ανάπτυξη. Ωστόσο, δεν είναι αυτός ο μόνος, η μόνη φιλοδοξία. Πρώτον, εσείς ως ε, άμεσα ερετή εκπρόσωποι αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι, παίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στον τομέα της ανάπτυξης. Στο, για το προσεχές λοιπόν δημοσιονομικό πλαίσιο προτείναμε το πρόγραμμα ενίσχυσης να διατηρηθεί και στην ε, πρόσφατη ανακοίνωσή μας για τους οργανισμούς ή τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών προβλέπονται και ειδικά κονδύλια. Επίσης, οι τοπικές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις βασικές ανάγκες των ε, πολιτών μέσω της αποκέντρωσης και της περιφερειακής προσέγγισης. Έτσι λοιπόν το προσεχές ε, έτος θα εγγενιάσουμε τη νέα εταιρική σχέση με τις ε, τοπικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση και τη συνεργασία με τις τοπικές διοικήσεις της αναπτυσσόμενες χώρες. Δεύτερον, όπως έχω επαναλάβει στο παρελθόν, η βιώσιμη γεωργία και η ασφάλεια των τροφίμων και της ε, διατροφής είναι θεμελιώδους σημασίας. Πρέπει να είμαστε το πρότυπο για τη συνεργασία ε, στο τομέα της βιωσιμότητας στη γεωργία. Μόνο μέσω αυτής της πολιτικής μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια άρρηκτη σχέση μεταξύ ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας. Έτσι λοιπόν, με την ανακοίνωση που θα κάνουμε στο θέμα αυτό το προσεχές έτος θα διασφαλίσουμε ώστε οι βέλτιστες τακτικές, πρακτικές να γίνουν ε, στάνταρ πρακτικές. Είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε την κοινή μας πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων και της ε, διατροφής ή της σύντησης. Απαιτείται συντονισμό των δράσεών μας. Θα σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του χρόνου. Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω την απόλυτη υπεποίθησή μου ότι θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσε αποτελεσματικά στη χορήγηση ανθρωπιστικής ε, βοήθειας ή βοήθειας στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας μέχρι τώρα και μέχρι το 2015. Από κοινού, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη της είναι ο μεγαλύτερος δωρητής του κόσμου που προσφέρει πάνω από το ίμιση της ε, αναπτυξιακής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και πολύ περισσότερο από τις ΗΠΑ. Επίσης, είμαστε και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος ε, των αναπτυσσόμενων χωρών και η μεγαλύτερη οικονομία που δίνει ελεύθερη πρόσβαση για... Που δίνει τη δυνατότητα οι χώρες αυτές να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην τροφή, στο καθαρό νερό. Και υποσχόμαστε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα θα συνεχίσουμε να πιέζουμε με αυτό το 0,7% που έχουμε δεσμευθεί, δεσμευθεί για το στόχο του 2030. Όλες οι χώρες μέλη, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες εποχές, μπορούν να αποδώσουν καλύτερα και να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα για αυτούς που χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας η φωνή τους δεν ακούγεται, αλλά βασίζονται σε εμά. Γι' αυτό λοιπόν κάνω έκκληση προς εσάς να με στηρίξετε και να με βοηθήσετε να μιλήσω και εξ ονόματός τους. Αυτή η υποστήριξη θα εκτιμηθεί ιδιαίτερος και ελπίζουμε ότι το 2013 θα είναι το το βέλτιστο έτος για όλους. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ευχηθώ χαρούμενα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Κόρτε Κάστρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ. Με μεγάλη χαρά ακούσαμε το πρόγραμμά σας που μας το παρουσιάσατε για το 2013. Θα ήθελα να μιλήσω καταρχάς για αυτά που είπατε εσείς και θα ήθελα να σας να σταθώ στις εξηγήσεις που μας δώσατε. Ελπίζω το Μάρτιο να σταθείτε περισσότερο, με περισσότερες εξηγήσει. Οι στόχοι ανάπτυξης της πολιτείας θα πρέπει να λάβουν υπόψη ε, την κατάσταση στην οποία ζούμε. Τις οικονομικές δυσχέρειες. Η πολιτική αυτή μέχρι το 2015, η πολιτική δηλαδή ε, αναπτυξιακής βοήθεια ε, είναι, αντιμετωπίζει κινδύνους. Ε, πρέπει να βρούμε και άλλους στόχους φιλόδοξους από το 2015 και μετά. Υπάρχουν τρία θέματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Καταρχάς, η δημοσιονομική υποστήριξη. Ε, υπάρχει αυτή η ανακοίνωση που πρόσφατα παρουσιάσατε Υπάρχει μια σειρά από κόκκινες γραμμές και το τελικό αποτέλεσμα είναι θετικό. Πολλές κυβερνήσεις ε, το αποτέλεσμα αυτό το υποδέχτηκαν θετικά. Είναι σίγουρο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουμε προσπάθειες ε, υποστήριξης των προϋπολογισμών πολλών ε, αναπτυσσόμενων χωρών. Αλλά είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τι γίνεται με τις χώρες όπου υπάρχει σημαντική διαφθορά. Θα ήθελα λοιπόν να στείλω ένα μήνυμα και να πω. Φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους εσωτερικούς ελέγχους και λυπάμαι που δεν έχουμε θεσπίσει ως κριτήριο την καλή διακυβέρνηση. Και θα ήθελα να σταθώ στο θέμα λίγο της ε, δημοσιονομικής ε, υποστήριξης και να κάνω ένα προβληματισμό. Ε, φυσικά μιλάμε πολύ για αυτό το θέμα προβάλλεται έτσι η αναπτυξιακή μας βοήθεια μέσω αυτής της στήριξης. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω αυτή τη δημοσιότητα που δίνουμε στην αναπτυξιακή μας βοήθεια. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία. Πρώτη σκέψη. Καταρχάς πώς εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Δεν υπάρχει σχέδιο εφαρμογής. Θα πρέπει αυτή να υπάρχει σε όλα τα νέα μέσα αναπτυξιακής βοήθειας. Και θα ε, τελειώσω με το συντονισμό των ε, συντονιστών. Ε, το είχαμε συζητήσει στην αρχή της θητείας μας, της κοινοβουλευτικής μας θητείας, αλλά δεν προχωρήσαμε πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή μας σύντομα θα κάνει μια νομοθετική πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη, θα κάνει μια πρόταση σύντομα Ποια είναι η άποψή σας για το συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και τη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πίμπαλξ για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε το πρόγραμμα και τις παρατηρήσεις που έκανε επί της ουσίας. Τέσσερα σημεία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Καταρχάς τη χρηματοδότηση. Σας ομολογώ ότι κάνουμε σημειωτών εδώ. Ε, και, και μάλιστα πολλά λέω, για να μην πω ότι παναχωρούμε. Ακούμε πάρα πολλά εδώ στο εσωτερικό της Επιτροπής και είχαμε και ανταλλαγή απόψεων με την Κύπρια Υπουργό Εξωτερικών εδώ πρόσφατα που ήρθε να μας παρουσιάσει τα θέματα που αφορούν και τα όσα κάνει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ήταν απογοητευτική αυτή η συνάντηση. Το μόνο που μας παρουσίασε ήταν την ανικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν τις δεσμεύσεις τους, τις υποχρεώσεις τους. Ως πολιτικό όργανο η Επιτροπή μας δεν μπορεί να τα δεχτεί αυτά. Πρέπει να αρχίσουμε να τραβάμε τα αυτιά των κακών κρατών μελών. Λέτε ότι χρειαζόμαστε πολύ έντονα επιχειρήματα για να πείσουμε τις δύσκολες χώρες. Πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή συνένεση για την ανάπτυξη. Έτσι. Και υπάρχει και υπογραφή για κάποιες δεσμεύσεις. Ε, δεσμεύσεις που θα έφταναν την οικονομική μας συνεισφορά στο 0,7%. Είχαμε δεσμευτεί για αυτό το 0,7%. Αυτό είναι ένα σημαντικό επιχείρημα. Το άλλο είναι το ηθικό επιχείρημα που το λέμε και το ξαναλέμε ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να εκριζώσουμε την φτώχεια. Τρίτο επιχείρημα. τι γίνεται μετά το τέλος της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει να υπάρχει εδώ η αρχή της διαφοροποίησης. Αυτή υπήρχε στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και η διάσκεψη του, της Νέας Υόρκης του φθινοπόρου του 2013 θα υπενθυμίσει σε όλους τους υπεύθυνου για την κρίζωση της φτώχειας, όχι μόνο στις χώρες δωρήτριες, αλλά και σε κάποιες από τις χώρες που είναι αποδέκτριες η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, ας πούμε, λέμε ότι δεν κάνουν αρκετά για να ξεριζώσουν τη φτώχεια. Ποιο στέει. Λέμε εμείς, ας πούμε, ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα πια για αυτή την ιστορία. Ε, είναι δικό τους θέμα πια. Θα πρέπει σε αυτή τη διάσκεψη της Νέας Υόρκης ε, αυτές οι χώρες να δεσμευτούν, ούτως ώστε οι δικές μας προσπάθειες μέσω από τις ε, αναπτυξιακή μα πολιτική να μην πάνε ει μάτιν. Τρίτον, αναφερθήκατε στι κατεξιοδότητε συμπράξει. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, που είναι να δώσουμε εξουσία απόφαση ίση με το Συμβούλιο στην Επιτροπή μας, σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά του στρατηγικού προσανατολισμού. σε ό,τι συνεισφέρει στο να πάρουμε αποφάσεις, πραγματικές πολιτικές αποφάσεις. Δεν ζητάμε κάτι το αδύνατο. Δεν, μιλάμε για μια μικροδιαχείριση εδώ πέρα, ε, διαχείριση δηλαδή από πολύ κοντά, με τρομερό έλεγχο και εκ του, σύνεχης, εκ του σύνεχης. Μιλάμε για την κάλυψη αυτού του δημοκρατικού α, ελλείμματος. Ε, 53 δισεκατομμύρια επιστρέφουμε το 80% από τα 53-54 εκατομμύρια πηγαίνει στα κράτη-μέλη. Το 10% πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. εκεί δεν έχουμε καθόλου λόγο. Στο 80% που δίνουμε στα κράτη-μέλη επίσης δεν έχουμε λόγο. Και το υπόλοιπο 10% ε, πηγαίνει στην, στο μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας. Και τα κράτη-μέλη σφίγγουν ακόμα περισσότερο το ζωνάρι, δηλαδή πιέζουν αυτό το 10% για να μειωθεί. Για αυτό το 10% θέλω να μιλήσω. Αν το κόψουμε κι άλλο. Ή αν θίξουμε την ε, εξουσία στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τότε θα φτάσουμε στο 5% της συνολικής βοήθειας για την ανάπτυξη από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ ντρέπομαι που αναγκάζεται η κοινή μας νόμη να δει αυτή την κατάσταση ότι παρουσιάζουμε αυτά τα πράγματα στον κόσμο μας. Πώς μπορούμε να εμφανιστούμε ψηλά το κεφάλι στους, εκλογείς, στους ε, ανθρώπους που μας ψηφίσουν και να τους λέμε ότι μπορούμε να επηρεάζουμε τα πράγματα. Όταν αυτό στο οποίο μπορούμε να πούμε θα το ξοδέψετε έτσι ή αλλιώς, σε αυτό το οποίο μπορούμε να έχουμε λόγο ας πούμε, είναι κάτω από το 10%. Είναι γύρω στο 5%. Από τα 53-54 δις, το 80% αφορά τα κράτη-μέλη, κανένα λόγο, το 10% επίσης δεν μπορούμε να το θίξουμε. Τώρα για το εμπόριο. Ε, διαπραγματευτήκαμε ε, εταιρικές σχέσεις οικονομικής φύσεως. Ο προκάτοχός σας ήθελε να εμπλακεί, αλλά του το απαγορεύσαμε. Σήμερα βρέπουμε τους καρπούς αυτής της αποτυχίας. Δηλαδή, ο Επίτροπος Ανάπτυξης από την αρχή δεν είναι, δεν από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Και έτσι επιλώνουμε πολύ ακριβά αυτή την καθυστέρηση ε, που είχαμε στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες ΑΚΕ. Τώρα είμαστε στη φάση επικύρωσης μιας συμφωνίας με τέσσερις χώρες ε, που είναι γελία οι υπόλοιπε 12 χώρε αυτή τη ε, γεωγραφική ομάδα γιατί δεν συμμετέχουν. Εσεί έχετε την υποστήριξή μα. Την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν ζητήσετε την αλληλεγγύη από τον κόσμο, από εμά, θα, σας θα τη δώσουμε για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει εσείς, μαζί με τον Επίτροπο που είναι υπεύθυνο για τα εμπορικά θέματα, να είσαστε πραγματικά στο ίδιο επίπεδο. Θα, έχετε, θα πρέπει να έχετε τι ίδιε εξουσίε, τι ίδιε αρμοδιότητε. Γιατί αλλιώ θα την πληρώσουν οι Αφρικανικέ χώρε και γενικά οι χώρε ΑΚΕ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα για την ανάπτυξη. Αυτή η περιφερειακή διάσταση μπορεί να δώσει μια νέα πνοή στην οικονομική ανάκαμψη αυτών των χωρών και κατά συνέπεια να τους δώσει τα μέσα για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θα ήθελα να μου απαντήσετε ειλικρινά. Και σας ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα ειλικρίνεια. Θα ήθελα όμως και άλλοι να πάρουν το λόγο. Κυρίως το Συμβούλιο, το οποίο μονίμως πει την ίσαν. Δεν λέει κουβέντα. για όλους τους τομείς για τους οποίους μίλησα θα πρέπει και αυτό να μιλήσει, το Συμβούλιο να μιλήσει. Θα πρέπει να σεβαστεί την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και να θεωρήσει ότι είμαστε ισότιμος εταίρος σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Είμαστε ισότιμος συνομοθέτης. Είμαστε ένας από τους πυλώνες μαζί με το Συμβούλιο ε, στη συνένεση που δημιουργείται για την αναπτυξιακή βοήθεια. Βασίζομαι σε εσά ούτω ώστε να ταράξετε λίγο τα λιμνάζοντα ύδατα. Επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια, αλλά ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Λέμε, ότι θέλουμε ισοτιμία σε νομοθετικό επίπεδο καμία συνέχεια δεν δίνεται. Επίση, λέμε, θέλουμε τα κράτη-μέλη να σέβονται την υπογραφή του. Δεν γίνεται τίποτα. Λέμε, θέλουμε περισσότερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και ημών. Καμία συνέπεια. Καμία συνέχεια. Αρχίζουμε να κουραζόμαστε και εκείνοι που κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν αποθαρρύνονται σε αυτή την ευγενή μάχη που είναι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα τον εαυτό μου, στον εαυτό μου το λόγο. Κύριε Επίτροπε, καταρχάς σας ευχαριστώ που είστε εδώ και που μας παρουσιάσατε το πρόγραμμα εργασίας σας για το 2013 στα πλαίσια του διερθωμένου διαλόγου. Προσυπογράφω απόλυτα αυτά που μόλις τώρα είπε ο συνάδελφος. Σας υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο και η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή εκπώνησε για σας δύο σημαντικά σημεία που θα ήθελα να ξαναβρει να υπάρχουν στο πρόγραμμα εργασίας σας. Τα ευρωπαϊκά γονδύλια σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελέσουν ένα project που να συνδέεται με κάποιον τρόπο με τα βιοκάψιμα και να χρησιμοποιούμε δηλαδή την αρωτρέα γη για να παράγουμε βιοκαύσιμα. Ποτέ δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Ε, εδώ ε, μιλάω για το πρόγραμμά σας για την επιστημιστική ασφάλεια. Αυτό είναι το ένα θέμα που θα ήθελα να υπάρχει. Το δεύτερο σημείο που θα πρέπει να απασχολεί στην Κομισιόν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συνέπεια των αναπτυξιακών μας πολιτικών με τις συμβάσεις που υπάρχουν ε, για, το ελεύθερο εμπόριο ή τις συμφωνίες για το ελεύθερο εμπόριο. Αυτά τα δύο σημεία που απασχολούν πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενυπάρχουν στο πρόγραμμα εργασίας σας του 2013. Η επόμενη ομιλήτρια. Äh, Ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους μου κύριε Επίτροπε θα ήθελα να δείξω το θέμα της πολιτικής συνέπειας. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα και αν δεν το αντιμετωπίσουμε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αναπτυξιακή πολιτική. Τα τελευταία δύο χρόνια όπου ήμουν συγγήτρια, τώρα ο κύριος Τσάλσε έχει την ε, χαρά να εξετάζει αυτό το τόσο δύσκολο θέμα. Εγώ λοιπόν έκανα την εξής εμπειρία. Υπάρχει μια σειρά επιτροπών που αδιαφορούν παντελώς για το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι θέμα δικό μας αλλά και της Επιτροπής. Το θέμα αυτό να το ε, προβάλλουμε περισσότερο, να συζητηθεί σε βάθος, διότι βέβαια ε, θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσουμε αν δεν το κάνουμε. Αν, ας πούμε, η Επιτροπή μπορεί δεν ασχολείται με τα θέματα αυτά, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Θα υπάρχουν συνεχώς ε, φραγμοί που θα τους έχουμε ανεγείρει μόνοι μας. Νομίζω λοιπόν ότι στον τομέα αυτό πρέπει να προβάλλουμε το θέμα και σας είπα τόσο η Επιτροπή όσο και οι βουλευτές. Να δείξουμε πόσο σημαντικός είναι ο τομέας αυτός. Και νομίζω ότι αυτό αναφέρεται και στην ε, έκθεση της Επιτροπής. Θα ήθελα να στήσω τον κύριο Charles Ντορίνγκ σχετικά με αυτά που είπε ε, στην εισήγησή του. Νομίζω ότι και εκείνος, όπως και οι άλλοι, ε, πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό τομέα. Δηλαδή, αν δεν καταρθώσουμε τις φτωχές χώρες να τις βοηθήσουμε να αναπτύσσουν μόνες τους εμπορικές συναλλαγές, να εισπράττουν φόρους από εκείνους ε, που φοροδιαφεύγουν, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εξαλείψουμε τη φτώχεια στις χώρες αυτές. Και πρέπει να σας πω, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όσο εσείς. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε αυτά μέχρι το 2013. Πάντως πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Και επιτρέψτε μου και μία τελευταία σκέψη, έτσι με λιγάκι επιφυλακτική ε, και εσείς το είπατε και χάρηκα ιδιαίτερα σχετικά με το, την άποψη ότι η Ευρώπη πρέπει να ομιλεί με μία και μόνο φωνή. Εγώ όμως σας είπα, είμαι επιφυλακτική. Υπάρχουν τόσες πολλές, πολλές φωνές που ακούγονται για διάφορα θέματα που δεν νομίζω ότι αυτό θα το καταφέρουμε γρήγορα και θα χαρώ πάρα πολύ αν η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μπορέσει να το πράξει αυτό και εν πάση περιπτώσει έστω εδώ ανάμεσά μας σας μιλάμε και με πολλές φωνές και τσακωνόμαστε κιόλα. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ε, ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις και για τις ερωτήσεις που μου υποβάλλατε θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που ελέγχεται προηγουμένως. Κοιτάξτε, υπάρχει πράγματι ένα οπλοστάσιο. Το θέμα είναι αν θα το χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Έχουμε κινητοποιήσει ε, περίπου ένα δις ε, για διάφορα εργαλεία που εντάσσονται στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Πάντως, οι προσπάθειές μας πρέπει να εστιαστούν ε, στην πρόθεση των στόχων αυτών, να ασκήσουμε μεγαλύτερη επιρροή. Τώρα, όσον αφορά τη μερίσια διάταξη μετά το 2015, έχουν ακουστεί διάφορες και διαφορετικές απόψεις. Για μένα, αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι ε, θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και οι στόχοι μας να είναι μετρήσιμοι. Γιατί αν σε τελική ανάλυση καταλήξουμε σε, ένα, σε μια μεγάλη βεντάλια, χωρίς ε, να μπορούμε να μετρήσουμε την επιτευχθήσα πρόοδο, νομίζω ότι τότε θα έχουμε χάσει την ευκαιρία. Γιατί η όλη δυναμική που χαρακτηρίζει τους στόχους χιλιετίας είναι αναμφίβολα θετική. Ας πούμε, στις συζητήσεις ε, για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο εξακολουθούμε να θεωρούμε το 0,7 ως ΑΕΠ ε, μέχρι το, του ΑΕΠ μέχρι το 2015. Αυτή λοιπόν η διάσταση των στόχων της χιλιετίας είναι τόσο σημαντική για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια που πρέπει να την προβάλλουμε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που ακολουθούμε και βεβαίως και ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικός σε αυτή τη διαδικασία μετά το 2015. Δεκυβεύονται πολλά θέματα Πάντως, αυτό που είναι το σημαντικότερο είναι να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια. Τώρα, όσον αφορά τη δημοσιονομική υποστήριξη, την στήριξη του προϋπολογισμού, ε, θα τεθούν κάποια θέματα. Πάντως, ε, υπήρξε μία πολύ ενδιαφέρουσα αξιολόγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας. Και τι διαπίστωσε. Διαπίστωσε μία σειρά σημαντικών θεμάτων. Πρώτον, λένε στο Υπουργείο Εξωτερικών της ότι υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στην στήριξη του προπολογισμού και την επίτευξη των στόχων χιλιετίας. Ξεκάθαρα το λένε αυτό. Δεύτερον, λένε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στην έγκριση του προπολογισμού και την αύξηση της διαφθοράς. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η έγκριση του προπολογισμού χρησιμοποιήθηκε ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Ούτε βέβαια και η φτώχεια μπορεί να επιτευχθεί. Αλλά εκείνο που παίζει ρόλο είναι ότι η έγκριση του προϋπολογισμού δεν σχετίζεται με την διαφθορά. Εμείς ε, πληρώνουμε περισσότερο με βάση την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων ε, την, ε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μερικές φορές φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου δεν επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. Το, 12, το 2011 δαπανήθηκε, εκταμιεύτηκε ένα μεγάλο ποσό με τη μορφή βοήθειας είναι σημαντικό να τηρούμε τις υποσχέσεις μας, γιατί αν δεν εκταμιεύουμε τα κονδύλια αυτό, πλήττει τους φτωχούς. Πάντως, ε, εκείνο που ενδιαφέρει είναι τα κονδύλια να μην ε, είναι αντικείμενο κατάχρηση. Κοιτάξτε, η μελέτη που έγινε κατέληξε στο ότι δεν μπορεί κανείς να αγοράσει πολιτικές μεταρρυθμίσεις με οικονομική βοήθεια με κονδύλια που εκταμιεύουμε. Υπήρχαν πολλές ε, προσδοκίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση, αλλά κατ' ουσίαν οι κυβερνήσεις ακολουθούν, εξακολουθούν, ακολουθούν το δικό τους το ρυθμό και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η οικονομική ενίσχυση που χορηγούμε ε, βοηθάει τις ε, χώρες που τη λαμβάνουν. Πάντως, η οικονομική ενίσχυση προσαρμόζεται και υπάρχει αυτή η οξελόγηση που σας είπα που έγινε και που επιβεβαιώνει ότι ε, έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα. Τώρα, όσον αφορά την κοινωνική προστασία και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, νομίζω ότι η ανακοίνωσή μας είχε καλή επίχυση. Εμείς ε, θέλω να πω το εξή. Όταν μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε καταρχήν για τους ανθρώπους που ζουν στην επαρχία και τα φτωχότερα στρώματα. Η ενίσχυση που δίδεται για την διατροφή αφορά κυρίως τους πιο φτωχούς, δηλαδή επουδενή δεν προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Και ε, σας είπα, η βοήθεια δίδεται στους ε, πιο φτωχούς. Σωστά είπατε ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή όχι της ε, σωστής πολιτικής. Και εγώ θα αναζητήσω στοιχεία και θα τα διαβιβάσω στον πρόεδρο της Επιτροπής να δούμε τι τελικά έγινε με αυτή την ανακοίνωση. Γιατί ε, πιστεύουμε ότι τα βήματα που γίνονται είναι σωστά. Τώρα, όσον αφορά το συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επ' αυτού θέλω να πω ότι υπήρξαν θετικές εξελίξεις. Και το πιο σημαντικό στοιχείο προέρχεται από τα κοινά προγράμματα. Δηλαδή αυτά τα οποία δεν είχαν απαραίτητα καλή επίχυση στα κράτη-μέλη. Θα θυμάστε ότι για κάποια προγράμματα συμμετείχαν πέντε χώρες, τώρα συμμετέχουν εννέα. Νομίζω όλο και περισσότερες χώρες αρχίζουν να ενθαρρύνονται, να θέλουν να συμμετέχουν σε εκείνα προγράμματα. Και αυτό σημαίνει ότι προσβλέπουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και κοινέ δράσεις, έτσι ώστε να, είναι, να χρησιμοποιείται ε, καλύτερα η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την ερώτηση του John Κάρλτ, θέλω να πω ότι η δική σας η χώρα, το Λουξεμβούργο, εξακολουθεί να τα καταφέρνει μια χαρά. Το ίδιο ισχύει και για την Δανία και για την ε, Σουηδία. Η Ολλανδία, κοιτάξτε, εκεί έγινε μια πολύ σκληρή συζήτηση, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το 0,7 και ελπίζω να παραμείνουν εκεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο κινείται προς το 0,7. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τη Φιλανδία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό το περίφημο negotiation box ε, να ε, καταλαμβάνει το 0,7% διότι από τη στιγμή που ε, θα αποθαρρυνθείτε, νομίζω τότε θα τελειώσουν τα πάντα. Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε στην ίδια κατεύθυνση γιατί έχουμε αρκετούς συμμάχους θα μπορούσα να αναφέρω, ας πούμε, την Ιταλία που τάχθηκε αναμφίβολα υπέρ της υποστήριξης του 0,7%. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση που το έχουμε υποσχεθεί. Ε, τώρα ζούμε μια δύσκολη εποχή και δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί να πρέπει να αποδεσμευτούμε από τις υποσχέσεις μας. Όσον αφορά τώρα αυτό το, την εκδήλωση το 2013, νομίζω ότι θα είναι μια κρίσιμη εκδήλωση σχετικά με τις εξελίξεις μετά το 2015. Γιατί τελικά, αν δεν είναι σαφές το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ε, δεν ξέρω, είναι δύσκολο όλο αυτό το εγχείρημα. Τώρα μεμονωμένες χώρες πρέπει να αναλάβουν υποχρώσεις, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ευρύτερος στόχος και οι μεμονωμένες χώρες πρέπει να εφαρμόζουν ε, προγράμματα ε, που εντάσσονται σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι οι χώρες πρέπει να ε, προσφέρουν ουσιαστικά, ουσιαστική βοήθεια στην εξάλληψη για την εξάλληψη της φτώχεια. Οι Κινέζοι και οι Ινδοί πρέπει να ενθαρρυνθούν ότι δηλαδή θα έρθουν οι κυβερνήσει τους και δεν θα τους αφήσουν να συνεχίσουν να ζουν στη φτώχεια. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία. Γι' αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα στο στόχο και μετά στα οικονομικά, όχι και τα δύο μαζί. Πρέπει ε, να υπάρχουν συγκεκριμένες φιλοδοξίες και στόχοι για κάθε χώρα. Τώρα, ως προς τις ε, Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Ε, υπάρχει μια πρόκληση να βρούμε την σωστή διατύπωση που θα επιτρέπει να υλοποιηθούν αυτά που είπατε και τελικά εγώ πάντα πίστευα ότι αυτή η Επιτροπή είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των φτωχών ανά τον κόσμο. Επίσης, ε, ε, θα πρέπει όμως να υπάρχει και ταχεία αποτελεσματικότητα όχι να μην ενστιάζουμε μόνο στο πνεύμα. Όσον αφορά στο εμπόριο, εδώ είμαι λιγάκι περισσότερο απεσιόδοξο σχετικά με το τι μπορούμε να πετύχουμε. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβάται την ε, πρόσβαση των ε, φτωχότερων χωρών στο εμπόριο. Σήμερα βλέπουμε ότι το θέμα προσεγγίζεται περιφερειακά και Δυστυχώς ε, οι προκλήσεις είναι διαφορετικές σε κάθε χώρα. Ας πάρουμε τη Δυτική Αφρική. Έχουμε την Γκάνα και έχουμε και το Τόγκο. Ε, δύο τελείως διαφορετικές οικονομίες. Είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίζει κανείς από κοινού και να συμφωνήσει για τα αποτελέσματα. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το σχέδιο που εφαρμόζεται είναι σωστό και το συνέλαβαν οι εταίροι μας. Ε, Βέβαια όσο περνάει ο χρόνο ε, η περιφερειακή ολοκλήρωση δεν είναι τόσο ισχυρή. Και όταν μιλάμε ε, σε πολιτικό επίπεδο, ε, εγώ έρχομαι από μια συνάντηση των ΑΚΕ και αυτό το πρόγραμμα το ΕΠΑΣ που είναι οικονομική εταιρική συνεργασία πραγματικά συζητήθηκε εκεί. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι δεν είναι το πρόγραμμα ΕΠΑ αυτό καθεαυτό περί οικονομικής ε, συνεργασίας που παίζει ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι το πώς εφαρμόζεται στις διάφορες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης θα συμμετέχει με μεγάλη χαρά σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εμείς συμμετέχουμε σε αναπτυξιακά κεφάλαια. Νομίζω όμως ότι τα αναπτυξιακά αυτά κεφάλαια δεν παίζουν άμεσο ρόλο στην Οικονομική Συμφωνία εταιρική σχέση. Η ε, συνάντηση κορυφή των ΑΚΕ με ανησύχησε λίγο γιατί εκεί τέθη ε, το θέμα από πολιτική σκοπιά. Ε, υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις χώρες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ, με πάση περιπτώσει, επιθυμώ να μειώσω την πολιτική χρειά σε τεχνικής φύσεως θέματα. Πάντως είναι προτεραιότητά μας. Η κυρία Ευαζολή ρώτησε για τα βιοκάψιμα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να προβλέψουμε κάτι συγκεκριμένο. Όσον αφορά συγκεκριμένα αυτό το θέμα, πιστεύω ότι η ανακοίνωση για τη διατροφή θα πρέπει να τύγει αυτό το θέμα. Η υπηρεσία μου πάντως έχει πει ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει κανένα πρόγραμμα σχετικά με τα βιοκαύσιμα. Να μην ασχοληθούμε με την τεχνική εξέλιξη στα βιοκάψιμα, ούτε καν με συμβιβασμούς. Ε, εκεί να μην αγγίξουμε καθόλου. Τώρα, όσον αφορά την συνδιάσκεψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ε, ε, Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών, αυτό είναι ένα θέμα που ετέθη με σαφήνεια και δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίφαση. Είναι σαφές ότι υπάρχει συνέπεια και συνέχεια. Αλλά αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, εγώ να σας ε, προσφέρω και άλλες εγγύησεις, διότι πιστεύω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί κανείς να τα πουλήσει. διότι το θέμα των μεμονωμένων ε, διαπραγματεύσεων. Μερικές φορές υπάρχουν βέβαια και τα εμπορικά μυστικά. Η ε, ανακοίνωση που παρουσιάστηκε εντάσσεται σε αυτό το πνεύμα. Σχετικά με την ερώτηση ε, της ειρήνης και της ανάπτυξης, κοιτάξτε, πράγματι οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι η ειδοποιώς διαφορά. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι αναφορές για κάθε συγκεκριμένο ε, project ε, βοηθούν στο να προχωρήσουμε γιατί με τον τρόπο αυτό μας προσφέρεται η ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε και εμπορικής ε, φύσης θέματα και θέματα εισοδημάτων. Η διαφάνεια λοιπόν ε, στον τομέα της επεξεργασίας ε, ξύλου και των εξορίξεων. Ε, αυτό είναι καθοριστική σημασία. Πρέπει να εστιάσουμε εκεί την προσοχή μας και στο μέλλον. Και υπάρχει και η Συμφωνία Λίας και αυτά είναι καλά και σημαντικά, αλλά πιστεύω ότι η διαφάνεια είναι το καθοριστικό στοιχείο. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη διαφάνεια είναι καθοριστική σημασίας. Έτσι λοιπόν σήμερα το διεθνές πλαίσιο έχει πολλά παραθυράκια, δυστυχώς ακόμα και είδα την έκθεση της ε, Προέδρου πριν από ε, λίγο καιρό. Ε, δυστυχώς δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση και ελπίζω να επικρατήσει διαφάνεια στην εξορρυκτική βιομηχανία αυτό θα είναι σημαντικό βήμα προς τα εμπρό, γιατί είναι αλήθεια ότι οι αναπτυσσόμενε χώρε έχουν πολλές διαρθρωτικές ε, αδυναμίες. Αλλά σας λέω, η πλήρη διαφάνεια είναι η απόλυτη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. Τώρα, στόχοι 2030, πολύ φιλόδοξοι, αλλά μην ξεχνάτε, μιλάμε για μετά από 18 χρόνια. Και αν τα παιδιά μέχρι και τότε δεν θα τρέφονται σωστά, τι να πω, ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακραία φτώχεια. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, ε, στην υγεία, στην κατοικία, αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε το να μιλάμε με μία φωνή. Αυτό οπωσδήποτε είναι μία πρόκληση. Ελπίζω μετά την ε, κατεύθυνση που θα δοθεί για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και την ολοκλήρωσή της, ίσως μπορέσουμε πράγματι να επιτύχουμε μεγαλύτερη συνέχεια και συνέπεια στην αναπτυξιακή πολιτική. Λυπάμαι που δεν υπάρχει στον τομέα αυτό κοινοτικό και εκτομένο. Πρέπει να υπάρξει ίσως την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Το θέμα δεν είναι πώς δαπανάμε σήμερα τα χρήματα. Δυστυχώς είμαστε πολύ διαρρεμένοι και πρέπει να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Σήμερα δουλεύουμε περισσότερο ευτελεντικά, εκεί υπάρχουν όρια. Σας είπα προηγουμένως, η δυναμική που χαρακτηρίζει τα κοινά προγράμματα είναι πολύ καλή. Όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αυτή δουλεύει καλά, άρχισε τώρα να εμπλέκεται σε διαδικασίες ε, προγραμματισμού Όλη αυτή η συζήτηση είναι πολύ σωστή, υγιής. Ε, η μία είναι πολιτική, η άλλη είναι πιο συγκεκριμένη και έχει σχέση με στόχους. Πάντως αυτό που παίζει ρόλο είναι να υπάρχει συνέπεια ε, στην ανάπτυξη και στην υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης. Στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης προσπαθούν να δουλεύουν με μεγαλύτερη συνέπεια με τα κράτη-μέλη. Ε, και αυτό, αυτό και για αυτές και για τα κράτη-μέλη είναι πρόκληση. Ε, πάντως, σε ορισμένες υπήρους τα πράγματα πάνε καλύτερα, σε άλλες πάλι ε, όχι τόσο καλά. Η δυναμική είναι αναμφίβολα καλύτερη και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε αυτό το στόχο του να μιλάμε με μία φωνή. Σήμερα Έχουμε πολλές δυσκολίες, αλλά εν πάση περιπτώσει ο αρμόδιος επίτροπος όταν μίλησε για την ολοκλήρωση οικονομικής και νομισματικής ένωσης είπε ότι πρέπει να μιλάμε με μία φωνή και είναι απόλυτα σαφώς ότι οι συνεισφορές μας ε, δεν είναι και όλες οι ε, ίδιες. Εγώ ε, θέλω να πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μία ρήξη μια τομή σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Το να μιλάμε με μια φωνή ε, και στο Διεθνές νομικό Ταμείο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Merci beaucoup. La parole est à monsieur. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γκέρνς. Merci comme la générosité. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχα... Ευχαριστώ πολύ για την γενοδορία ε, από πλευρά του Επιτρόπου. Θα ήθελα κύριε Βίμπεξ να, έρθω στο θέμα, να επανέλθω στο θέμα του εμπορίου. Ε, μας δίνεται ένα επιχείρημα, επιπρόσθετο επιχείρημα, όχι μόνο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις μόνον, αλλά επίσης για να γίνουμε ηγέτες σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Γιατί με την ε, περιεκτική ανάπτυξη, ας πούμε, είναι προφανές ότι η ανάπτυξη έχει νόημα παρά μόνον έχει νόημα μόνο όταν συμβάλλει στην εξάλληψη της φτώχειας. Η ανάπτυξη λοιπόν η οποία ε, θα εξασφαλιστεί μέσω του εμπορίου θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτή η περιεκτική ανάπτυξη. Και στις διαπραγματεύσεις ο αρμόδιος ε, για το εμπόριο επίτροπος για τεχνικούς λόγους θα πρέπει να συμφωνήσει επί των πτυχών που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αλλά ως προς την ουσία, εσείς πρέπει να διαδραματίσετε το σπουδαιότερο ε, ρόλο, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια επιτυχώς. Δεύτερον, όσον αφορά το ποσοστό 0,7%. Το αναφέρουμε καθημερινά. Και πρέπει να ε, σκεφτούμε μία μέθοδο για να κινητοποιήσουμε τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν κάνουν τίποτα. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που ε, κάνουν αυτό που πρέπει. Από την άλλη υπάρχουν οι χώρες οι οποίες πλήττονται από την κρίση όπως και οι άλλες. Ε, αυτές οι οποίες όμως υπαναχωρούν, ε, που δεν κάνουν αυτό που πρέπει και Βεβαίω στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξαιρέσουμε την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και δεν πρέπει να απαιτούμε τίποτα από αυτήν. Υπάρχουν άλλε χώρε όμω που αντιμετωπίζουν σοβαρέ δυσκολίε. Ωστόσο, μεταξύ αυτών που υπαναχωρούν, υπάρχουν χώρε οι οποίε θα μπορούσαν θαυμάσια να κάνουν αυτό που υποχρεούνται. Ε, δεν θέλω να προκαλέσω δυσφορία σε εκπροσώπους αυτών των χωρών. Θα μπορούσαν θαυμάσια όμως να πράξουν την αποστολή τους. Αυτές οι χώρες λοιπόν θα πρέπει να κληθούν να μας πούν για ποιο λόγο δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Το, κάνουν σε άλλους τομείς, το κάνουμε σε άλλους τομείς, παραδείγματος χάρη στο τομέα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπου το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο ε, καλεί τον Υπουργό Οικονομικών των χωρών τους υπουργού οικονομικών των χωρών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως προς την δημοσιονομική πειθαρχία να έρθουν και να λογοδοτήσουν ανώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έλεγα λοιπόν ότι και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει λογοδοσία ανώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι από τη σκοπιά της δημοσιονομικής τεχνικής βλέπουμε πολύ καλά τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι το 2015. Ε, δηλαδή βαθμιαία και σταδιακά αυτή η επιβράδυνση θα συσσωρευτεί εις βάρος της υλοποίησης των στόχων μέχρι το 2015 και μετά το 2015. Πρέπει να κληθούν λοιπόν να μας πούν αν θέλουν να σεβαστούν και να τηρήσουν αυτούς τους στόχους. Αν δεν μπορούν να μας πούν πότε θα είναι σε θέση να τους τηρήσουν. Είδω λοιπόν κάποιες προτάσεις. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει απλώς να ε, παραμείνουμε αδρανείς και απλώς να κάνουμε την διαπίστωση της αδυναμίας και μόνον. Νομίζω ότι είναι καθήκον της δικής μας Επιτροπής αυτό. Αν βρούμε λοιπόν ικανοποιητικέ απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα είναι ήδη κάτι σημαντικό. Ε, και βεβαίω, αν παραμείνετε μέχρι τις 5 η ώρα είμαι βέβαιος ότι δεν θα ε, μετανιώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ Τσάρλς, είναι πάντα πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο να ακούω τις απόψεις σου ε, και του συναδέλφου Κάρολ, γιατί η δική του δουλειά είναι να διαπραγματευτεί και είμαι βέβαιος ότι θα το πράξει και θα τον βοηθήσω και θα τον υποστηρίξω και θα υποστηρίξω τις πρωτοβουλίες του για να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα για τους εταίρους μας. Σχετικά με το 0,7. Νομίζω ότι ο χρόνος περνάει και τώρα πια βρισκόμαστε προς το τέλος των διαπραγματεύσεων και πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Διότι πραγματικά η Ευρώπη έχει δεσμευθεί με το 0,7 και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για καμία χώρα να αποσυρθεί. Ακόμα και για την Ελλάδα που είναι μια διαφορετική περίπτωση όπως αναφέρατε. Ωραία, κάθε χώρα θα έχει ένα ε, αξιόπιστο, σχέδιο για να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της. Δεν είναι τίποτα το 0,7. Είναι αληθές ότι για κάποιες χώρες θα είναι δυσκολότερο να το επιτύχουν, αλλά είναι ευκταίος αυτός ο στόχος. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση σε κάθε μία χώρα ώστε να ε, υλοποιήσουν, να πραγματοποιήσουν τη δέσμευσή τους όλες οι χώρες. Δηλαδή, ονοματίζοντας και ε, χώρες δεν βγαίνει τίποτα. Όλες οι χώρες έχουν δυσκολίες. Κάποιες μεγαλύτερες δυσκολίες, κάποιες μικρότερες. Και εμείς έχουμε δυσκολία. Αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί ως προς το 0,7 και εμείς ως Κομισιόν θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να πιέσουμε τις χώρες. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, αυτή η Επιτροπή είναι η Επιτροπή η οποία πραγματικά ηγείται της προσπάθειας για τη στήριξη των φτωχοτέρων. Και ε, πιστεύω ακράδαντα ότι η δική μου επιτυχία το προσεχές ε, έτος εξαρτάται απόλυτα από την καλή συνεργασία με τη δική σας Επιτροπή και τη στήριξη της Επιτροπής σας ε, τη συνεργασία μεταξύ ημών και της γραμματείας και των δικών μου υπηρεσιών. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε οπωσδήποτε το 2013 να είναι ένα καλό έτος, ακόμη καλύτερο και από το 2012. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γκέρενς, μια και δεν είναι ακόμα πέντε η ώρα, ας ξαναπάρω το λόγο. Για να μιλήσω για αυτό το διαβόητο 0,7%. Με την κλασική σας ευγένεια, τελικά δεν φύγετε καθόλου τις χώρες τις οποίες θεωρώ υπεύθυνε για αυτή την αποτυχία. Και λέτε δεν πρέπει να στυλιτεύσουμε τους υπεύθυνου. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν θέλω να στιγματίσουμε γενικά τις χώρες, αλλά θέλω όμως να προχωρήσουμε βαθμιδών. Στην πρώτη φάση σας παρακαλώ να υποδείξετε τους υπεύθυνου των χωρών που κατηγορούν άλλους που δεν δεσμεύονται, που δεν σέβονται μάλλον τις δεσμεύσεις τους για την βοήθεια. Νομίζω ότι τα είπα όλα ξεκάθαρα. Υπάρχει μία χώρα η οποία τα πάει πολύ καλά, που βγήκε καλά από την κρίση και που υποδεικνύει τους άλλους που δεν τα καταφέρνουν και αυτή η χώρα όμως δεν, δεσμεύε, δεν ε, υλοποιεί το στόχο της ε, που είναι το 0,7%. Αυτή η χώρα θα πρέπει να την καταγγείλουμε. Αν ξεκινήσουμε έτσι, μπορεί να αλλάξουν γνώμη και άλλες χώρες. Ούτως ώστε να φτάσουμε πιο κοντά στο μέσο όρο ε, που θέλουμε να πετύχουμε από τώρα μέχρι το 2015. Και αν έχετε δυσκολίες, έχετε τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή να σας στηρίζει. Ε, πολλά, τέλος πάντων, για να μην πω όλοι, πολλά μέλη της ε, Επιτροπής ΔΕΔΕ. Αν έχετε δυσκολίες, μην διστάσετε να ζητήσετε τη στήριξή μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν χρειαστεί μάλιστα, είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε μία διάσκεψη ή μία νέα συνεδρίαση της Επιτροπής. Κύριε Επίτροπε, δεν θα είστε μόνος σε αυτόν τον αγώνα. Έχετε το υπόψη σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόρτες Λαστράς. Έχει το λόγο. Καταρχάς, ένα προβληματισμό για αυτές τις χώρες που πήραν μια σαφή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά είναι αυτές οι χώρες οι οποίες επηρεάστηκαν από την κρίση και τελικά μείωσαν το, τα κονδύλια για την ε, διεθνή συνεργασία. Ας πούμε η Ισπανία. Εμείς είχαμε μια σαφή ε, πορεία σε ό,τι αφορά την διεθνή συνεργασία, αλλά τελευταία ε, υπήρξαν δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό της αναπτυξιακής βοήθειας. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτών των περικοπών που είναι πολύ σημαντικό γιατί εγκαταλείπουμε προγράμματα και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γκέρενς. Κάποιοι υπεύθυνοι θα πρέπει εδώ να έρθουν και να μας εξηγήσουν, να λογοδοτήσουν γιατί αποφάσισαν να προβούν σε αυτές τις περικοπές στον προϋπολογισμό της αλληλεγγύης. Όλος ο τομέας της αλληλεγγύης, γιατί είναι πολύ υποτομής, όλη αυτή, όλος αυτός ο τομέας γενικά ε, έχει πληγεί. Ε, επίσης, ε, η κοινωνία των πολιτών αυτών των χωρών που λάμβαναν τη βοήθεια, επίσης πλήττεται. Κάνετε ένα προβληματισμό πολύ ενδιαφέροντα στην αρχή. Δεν ήθελα να το υπογραμμίσω περαιτέρω, γιατί μου φάνηκε πολύ καθαρό αυτό που είπατε. Η κοινωνία των πολιτών και στους στόχους της χιλιετίας και σε άλλους στόχους ε, που προωθούμε θα πρέπει να ζητάμε μια μεγαλύτερη συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών. Της κοινωνίας των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό η πολιτική συνεργασίας να είναι πιο ανοιχτή στην κοινωνία των πολιτών η αποκεντρωμένη συνεργασία. Αυτό είναι ένα τρόπο για να τα καταφέρουμε. Ξέρετε ότι στη χώρα μου ότι η αποκεντρωμένη συνεργασία είναι ένα σημαντικό τμήμα τη ε, συνεργασία εν γέννη. Η οποία όμω σχεδόν εξαφανίστηκε. Τέλο πάντων, μην είναι υπερβολικό, αλλά περίπου έτσι έγινε. Σύντομα, η Επιτροπή των Περιφερειών και άλλες οργανώσεις θα οργανώσουν διασκέψεις για τον ρόλο της αποκεντρωμένης συνεργασίας. Εσείς μιλήσατε για μια πιο εκ του συνεργασία, η οποία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εμπέδωση της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μέλλον, αυτή η αποκεντρωμένη συνεργασία τι ρόλο πρέπει να παίξει Πώς θα τα καταφέρουμε τόσο ώστε οι χώρες που πλήττονται από την κρίση να υποφεληθούν. Μετά την πρώτη μου παρέμβαση έχω διάφορες ανησυχίες. Ε, ξέρετε ότι η πολιτική μου ομάδα θέλει δημοσιονομική στήριξη. Τη θέλει αυτή την πολιτική. Θεωρούμε ότι έχει δώσει καρπούς και θέλουμε να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά τους στόχους ανάπτυξης ε, της χιλιετίας, αλλά θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστές παράλληλα. Δεν θέλω να φτάσουμε στο 2015 και να κουβαλάμε ακόμα τις συνέπειες της κρίσης. Μια κρίση που μας έχει επηρεάσει όλους. Τέλος. Κλείνοντα, θέλω ακόμα να σταθώ στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να την ενισχύσουμε, αυτή την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει αυτές οι αξίες της αλληλεγγύη ε, στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκής Ένωση να τις ε, διδαχθούν, να τις μάθουν όλοι. Μέχρι τις 5 ε, η ώρα, κύριε Επίτροπε, έχετε ξανά το λόγο. Μάλιστα. Αυτά που μου είπατε ε, τα λάβαμε πολύ σοβαρά. Θα, στην έκθεση λογοδοσίας θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη μου αυτά που είπατε. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα και ξέρετε ότι οι διάφορε χώρε ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία, αλλά σίγουρα θα πρέπει να δούμε πώ αυτή η έκθεση λογοδοσία θα είναι αποτελεσματική και να είναι και πραγματικό έτσι εργαλείο. Τι αντιλαμβάνεται το κοινό τώρα. σε καιρό κρίσης όλοι μιλάνε για το ΑΕΠ. Υπάρχει μια σημαντική μελέτη από ένα think tank. για αυτό το θέμα. Στο, στη σημερινής στο σημερινό πλαίσιο για τις οικονομικές διαπραγματεύσεις, Ε, λέμε ότι η συμμετοχή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι σημαντική και όταν, όταν επενδύουμε στις, στις αντισόμενες χώρες, αυτό σημαίνει ανάπτυξη τελικά που έρχεται σε εμάς πίσω αυτό το 0,7% δεν, είναι μόνο, δεν γίνεται μόνο για την αλληλεγγύη, είναι επένδυση και για το δικό μας μέλλον. Νομίζω ότι αυτά τα επιχειρήματα θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Ε, να χρησιμοποιούμε παραδοσιακά δηλαδή οικονομικά επιχειρήματα για την αποκεντρωμένη συνεργασία. Πιστεύω ότι η ανακοίνωσή μας και οι προσπάθειές μας θα προωθήσουν και θα κρατήσουν ζωντανή αυτή την τάση. Τώρα, για τη στήριξη του προπολογισμού. το 2011 ε, το 18% ε, της βοήθειας πήγαινε ακριβώς σε τέτοια προγράμματα. Ο στόχος είναι να έχουμε μια κοινωνία χωρίς στόχια. Υπάρχουν, υπάρχει ένα εργοστάσιο α, το οποίο χτίστηκε από Νορβηγούς. Ε, χτίστηκε αλλά έμεινε τελικά χωρίς ενέργεια. Ποτέ δεν λειτουργήσε. Αυτά τα λεφτά ασπαταλήθηκαν. Αποκλείεται να ξαναλειτουργήσει. Απλώς θα μαραζώσει. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις για να προσπαθήσουν αυτές, για να προωθήσουν προγράμματα τα οποία θα εξαλείψουν τη φτώχεια. Πιστεύω ότι με προγράμματα υπέρ του περιβάλλοντος, υπέρ της ε, βιοπικιλότητας, ε, κάνουμε επενδύσεις ούτως ώστε να προωθήσουμε αυτό το στόχο της ε, εξάλληψης της φτώχειας. Ε, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε μέσω της στήριξης, της άμεσης στήριξης του προπολογισμού των αναπτυσσόμενων χωρών. Δεν κάνουμε μία μονόπαντη προσπάθεια. Πρέπει να κάνουμε παράλληλα προσπάθεια και σε, άλλες, σε άλλα επίπεδα, στο περιβάλλον, στην ενέργεια κτλ. Το θέμα είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. φτάνουμε στις 5 και θα τελειώσει εδώ η σχέση μας με τον... η συνομιλία μας με τον ε, Επίτροπο. Η ομάδα μου ήταν υπέρ του φόρου των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όταν θα υπάρχει αυτός ο φόρος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τμήμα από τα έσοδα για την εξάλληψη της στόχιας, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και για τη διεθνή συνεργασία. Χρήσιμο θα ήταν αυτό. Φυσικά, εγώ για το 0,7% είμαι πραγματικά θειασότης. Αλλά θα ήθελα να ασκήσουμε πιέσεις, ούτως ώστε να δουλέψουμε και σε άλλα επίπεδα. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνεται στο μέλλον αυτός ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Λοιπόν, νομίζω ότι η δέσμευση Νομίζω ότι η υλοποίηση του στόχου 0,7% ε, του 0,7% δέσμευση που πήραμε πριν από πάρα πολύ καιρό πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί. Οποιαδήποτε απόκληση θα είναι χαμένος κόπος. Βεβαίως πάντα υπάρχει αυτό το όνειρο του να υπάρξει αυτός ο φόρος κλπ. Αλλά η καταπολέμηση της φτώχειας ε, είναι ένα πραγματικό ε, γεγονός πραγματικό συμβάν. Θα ήταν ε, καλή προσέγγιση ένα μέρος αυτού του εσόδου, των εσόδων από το φόρο Επιχρηματοοικονομικών συναλλαγών να αφιερωθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας. Αλλά σήμερα βλέπουμε ότι κάποιες χώρες ε, θα, ήδη θα αρχίσουν να εφαρμόζουν αυτή τη φορολόγηση. Κάποιες χώρες όπως η Γαλλία, παραδείγματο χάρη, διαθέτουν ήδη το 10% για την ανάπτυξη. Δεν είναι αρκετό αυτό. Αλλά πάντως είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Και μας δίνει και θάρρος να σκεφτούμε ότι είναι ευκταίος αυτός ο, ο στόχος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις όπως είναι η φτώχεια, όπως είναι η αηφορία, η βιωσιμότητα και ίσως θα φτάσουμε σε κάποια φάση όπου θα μπορούμε να ε, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στη ρίζα τους. Κλιματική αλλαγή, παραδείγματος χάρη. Απαιτεί τεράστια χρηματοδότηση. Α, χρηματοδότηση του αναπτυσσόμενου κόσμου. Και ο ανεπτυγμένος κόσμος δεν, δεν έχει κάνει όσα έπρεπε να κάνει στο θέμα αυτό. και πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες αναπτυγμένες. Και βεβαίως η λύση ε, χρηματοδότησης από το φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ίσως είναι μια λύση αλλά στο απότερο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε που μοιραστήκατε μαζί μας ε, τους στόχους σας για το προσεχές έτος. Να γνωρίζετε βεβαίως ότι μπορείτε να βασίζεστε στην συνεργασία αλλά και στην εγρήγορση που επιδεικνύει η Επιτροπή μας σε θέματα ε, ανάπτυξης και με την ευκαιρία αυτή σας εύχομαι καλές διακοπές και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ Ξαναρχίζουμε. Πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης που αφορά την αλληλευτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας που καθορίζει τις αλληλευτικές δυνατότητες και το οικονομικό αντιστάθμισμα που προβλέπει η Συμφωνία εταιρική Σχέσης ε, για τα Αλληλευτικά που ισχύει ανάμεσα στα δύο μέρη. Η Επιτροπή μας γνωμοδοτεί απλώς. Η Επιτροπή Αλίας είναι η καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή φυσικά. Και ο εισηγητής μας, η εισηγήτριά μας μάλλον για τη γνωμοδότηση, η κυρία Γκεζίν Μεσνέρ, στην οποία δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, συγγνώμη που καθυστέρησα και με περιμένατε, αλλά ξέρετε εγώ είμαι και συντονίστρια σε μια άλλη επιτροπή ε, και είχαμε μια φλέγουσα συνεδρίαση και γι' αυτό λοιπόν έπρεπε δυστυχώς να παραμείνω λίγο εκεί και μετά να έρθω εδώ. Πάμε τώρα στη Μαυριτανία. Ε, από αναπτυξιακή σκοπιά η Μαυριτανία είναι μια χώρα με πολύ περιορισμένη ανάπτυξη, άρα δηλαδή εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το που ισχύει είναι το εξής. Η κυβέρνηση είναι ασταθής, αλλά έχει έναν ε, εκλεγμένο πρόεδρο. Η Αλκάιντα βέβαια ε, δραστηριοποιείται στη χώρα αυτή. Η τρομοκρατία είναι διαδεδομένη. Ε, κατόπιν τούτου για όλου αυτού τους λόγου χρειάζεται μια οικονομική σταθερή βάση. Ασχολείται με τη γεωργία στην χώρα, είναι δεδομένη η γεωργία και όσον αφορά τι εξαγωγές, εξάγονται ψάρια και ε, μέταλλα. Η χώρα είναι φτωχή, αλλά στην ακτή, μπροστά στην ακτή, αναπτύσσεται ελεία. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται τώρα και αυτή η συζήτηση. Περίπου το 50% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμφωνίες με ε, τρίτες χώρες και εταιρικέ σχέσεις αφορούν τη Μαυριτανία. Μιλάμε για 70 εκατομμύρια ευρώ και ε, εδώ ε, διακυβεύονται πολύ σημαντικά αλληλευτικά συμφέροντα ευρωπαϊκών κρατών. Προφανώς, ε, εμά δεν μα ενδιαφέρουν τα αλληλευτικά συμφέροντα, εμά μας ενδιαφέρουν τα αναπτυξιακά. Υπάρχει ήδη μία συμφωνία ανάμεσα Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαυριτανία που τέσσερι ισχύ το 2006. Υπήρξαν δύο συμπληρωματικά πρωτόκολλα και τον Ιούλιο ξέπνευσαν και αυτά. Έκτοτε έχουμε μια προσωρινή συμφωνία, η οποία όμως ε, καταλήγει και αυτή το 2013. Άρα δηλαδή ε, αυτή τη στιγμή μπορούν προσωρινά να υποβάλλονται αιτήσει και κατά κανόνα βέβαια εγκρίνονται. Το νέο πρωτόκολλο το οποίο έχει επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ισχύσει για δύο χρόνια από την ώρα που θα υπογραφεί. Η άλλη συμφωνία, όπως ε, σας είπα, εκπνέει τέλος του Ιανουαρίου, άρα δηλαδή πιεζόμαστε χρονικά να κάνουμε κάτι το υποσυζήτηση πρωτόκολλο διασφαλίζει ε, την πρόσβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλεονάσματα των αποθεμάτων. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Μαυριτανία ασκείται υπεραλίευση. Γι' αυτό λοιπόν το πλεόνασμα αυτό ε, δύναται να το αλλιεύει και να το λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό καλύπτει και τα ληφτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι αυτό εντάσσεται και μέσα στην βιώσιμη αλία. Μιλάμε λοιπόν για 70 εκατομμύρια ευρώ. 67 θα πάρει η Μαυριτανία, περισσότερα δηλαδή από ό,τι μέχρι τώρα, για να μπορούν οι ευρωπαϊκοί στόλοι να διεισδύουν στην ε, ζώνη αποκλειστική οικονομική εκμετάλλευση τη Μαυριτανία και τα υπόλοιπα 3 εκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν για την διασφάλιση τη βιώσιμη βιώσιμης αλίας. Αυτή λοιπόν η υποστήριξη της βιώσιμης αλίας παλαιότερα είχαν πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση, 20 εκατομμύρια τότε. Όμως δεν τα χρησιμοποιούσαν και αυτό τώρα υπήρξε μια ανακατανομή στη χρηματοδότηση. Σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες αλίευσης. Σας είπα, ένας λόγος είναι η υπεραλίευση. Ένας άλλος είναι ότι θα πρέπει και η Μαυριτανοί αλληλείς μόνοι τους να ασχολούνται με τη διαχείριση των αληφτικών τους αποθεμάτων. Και πάλι εδώ ε, υπάρχουν ε, διστάμενες απόψεις και ε, συγκρόμενα συμφέροντα, γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα της Επιτροπής Αλίας, της δικής μας και της Επιτροπής Γεωργίας. Οι Μαυριτανοί τα πήγανε πάρα πολύ καλά στις διαπραγματεύσεις και είπαν επίσης ότι τα κεφαλόποδα Φαντάζομαι ότι εδώ ε, δεν θα κάθονται ε, εμπειρογνώμες. Θα τολμήσω να πω, λέει ο Μιλήτρια, ότι αυτά είναι τα χταπόδια και κάτι άλλα. Αυτά εξαιρούνται, γιατί είπαν ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά για τους Ισπανούς. Και έτσι λοιπόν οι ε, γηγενείς αλληλείς επιθυμούν να διατηρήσουν αυτά τα κεφαλόποδα. Κεφαλόψαρα, με συγχωρείτε. Πρέπει λοιπόν να πούμε κεφαλόποντα. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε κατά πόσον υπάρχουν και ε, κινέζικα σκάφη ε, τα οποία επιθυμούν να λιεύουν εκεί στην περιοχή. Αυτό όμως δεν το επιθυμούν οι Μαυριτανοί. Ε, σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία παρότι από πλευράς αλίας, αλληλευτικής πολιτικής ε, για μας ε, έχει πιο δυσμενείς συνέπειες από ό,τι κατά το παρελθόν. Τώρα λοιπόν οι εφοπλιστές οφείλουν να συμμετέχουν αναλογικά οποτεδήποτε αλλιεύουν τα χωρικά ύδατα αυτά της Μαυριτανίας. Και επίσης, μόνο αυτό, εφόσον το πράττουν, να προσλαμβάνουν και Μαυριτανούς ε, ε, προσωπικό ως Μαυριτανούς. Εξαιρούνται τα κεφαλόποδα, το είπαμε αυτό. Η ζώνη οικονομικής αποκλειστικής εκμετάλλευσης επεκτείνεται στα 20 μίλια. Και αυτό ε, διότι κατά την αλλιεύση, αλλιεύονται και ψάρια τα οποία δεν τα ήθελαν οι Ευρωπαίοι, τα πετούσαν στη θάλασσα, τα θέλουν όμως οι Μαυριτανοί, τα καταναλώνουν αυτοί. Από πλευράς πολιτικής και οικονομικής όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί ενισχύουν ε, την ε, τοπική, το τοπικό εργατικό δυναμικό και εξάλλου ε, συμβαδίζουν και το, με τις δικές μας απόψεις για μια ολοκληρωμένη συμφωνία, κάτι το οποίο ήδη έχουμε εγκρίνει κατά το παρελθόν. Και υπάρχει και μια εξωτερική διάσταση στην κοινή αλληλεπτική πολιτική. Εξωτερική διάσταση γιατί, γιατί πρόκειται για μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα. Και κάτι άλλο. Το καλοκαίρι ε, συνήφθη μια συμφωνία για την ε, αλία στη Μαυριτανία, μια συμφωνία την οποία υποστήριξαν όλες οι πολιτικές ομάδες. Μακρηγόρησα, διότι ήθελα να σας εξηγήσω εξηγήσω ότι στην Επιτροπή Ελίας ε, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, αλλά από τη σκοπιά τη δική μας, την αναπτυξιακή, πρέπει να πω ότι πρόκειται για μια πολύ καλή συμφωνία. Κυρία Γκρέσ, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ και καλησπέρα. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος της Ελιζαμπέλα Λοβίνκη που είναι η εμπειρογνώμονάς μας για θέματα Ελίας, και μετά θα μιλήσω εξ ονόματος της ομάδας μου. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ την κυρία Μέσνερ για τη θαυμάσια έκθεσή της. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι με αυτή την ε, συμφωνία με τη Μαυριτανία μιλάμε για την πιο σημαντική ε, συμφωνία με τρίτη χώρα. Έχουμε πολύ θετική στάση για τις αλλαγές που υπάρχουν στη, στο νέο πρωτόκολλο. Αυτό το νέο πρωτόκολλο δεν επιτρέπει την πρόσβαση της, του ευρωπαϊκού στόλου ε, στα κεφαλόποδα, όπως υπενθύμησε η συγγήτρια. Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το αίτημα ήταν και αίτημα των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των μικρών αλλιέων της Μαυριτανίας, που εδώ και 10 χρόνια είχαν πρόβλημα ε, και πλήττονταν από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Επλήττονταν σε ό,τι αφορά την αλληλεία στα κεφαλόποδα. Χαιρόμαστε λοιπόν και γιατί αυτό το κείμενο που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ συνεπές σε σχέση με, τα, με όλα όσα ψηφίσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Παραδείγματος χάρη το ψήφισμα του Μαΐου του 2011 που έλεγε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Στόλου παρά μόνο στην αλληλεία ειδών ε, τα οποία δεν ψαρεύει ο στόλος της Μαυριτανίας. Επίσης, ε, αυτό το πρωτόκολλο είναι συνεπές και με την ε, έκθεση της Ιζαμπέλα Λοβίν για την εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, που έλεγε ότι ο Ευρωπαϊκός στόλος δεν πρέπει να ανταγωνίζεται τους μικρούς στόλους των εν λόγω χωρών, των, τους μικρούς δηλαδή ντόπιου αλληλείς. Για τα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ την προσοχή αγαπητοί συνάδελφοι στο γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και οι εκπρόσωποι των μικρών αλλιέων τη ε, Μαυριτανία συνεδρίασαν μέσα Οκτωβρίου για να συζητήσουν αυτό το νέο πρωτόκολλο. Το βρήκαν πολύ θετικό. Η σύστασή του είναι να μην ξανανοίξουμε τι διαπραγματεύσει Συμπερασματικά. Υπενθυμίσω το άρθρο 5 του νέου πρωτοκόλλου, το οποίο ζητάει τις ίδιες απαιτήσει που βαραίνουν το δικό μας στόλο να τις επιβάλλουμε και στους άλλους ξένους στόλους. Θα μπορούσε δηλαδή το πρωτόκολλο αυτό να αποτελέσει ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο ε, στις ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχετε λοιπόν την αμέριστη υποστήριξή μας, κύριε Συγγήτρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος, ο Νόισερ. Vielen Dank, Frau Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια την κυρία Μάισνα. Νομίζω ε, έχουμε μια συμφωνία λίες, ε, που είναι υποδειγματική, είναι καταπληκτική. Καταρχήν λοιπόν υπάρχει μια συμφωνία όπου εμείς ε, ως Κοινοβούλιο μπορέσαμε να επιβάλλουμε τα αιτήματά μας ε, που υποβάλαμε το 2011. Τα αιτήματά μας τα περάσαμε στο ψήφισμά μας. Ε, αυτή λοιπόν η συμφωνία Λίας με τη Μαυριτανία είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να μιμηθούμε στο μέλλον. Γιατί? Διότι πρώτον λαμβάνουμε υπόψη μας τα συμφέροντα των ντόπιων αλλιέων. Δεύτερον, ε, λαμβάνουμε υπόψη μας ε, την υπεραλήψη και επιθυμούμε να μην υπάρξει εξάντληση αλληλευτικών αποθεμάτων. Άρα δηλαδή να υπάρχει μια βιώσιμη αλληλευτική πολιτική. Η μεγάλη αλληλευτική στόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δυνατόν να ανταγωνίζονται τους ντόπιου αλληλείς και η μη κυβερνητική ε, οργανισμοί στην ε, Μαυριτανία, εφόσον αυτοί εγκρίνουν τη συμφωνία, καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ε, περικοπές ε, σε αυτή τη συμφωνία και έχουν νόημα αυτές, διότι τα αλληλευτικά αποθέματα ε, που την χάνουν υπεραλήψεις θα πρέπει να προστατεύονται. Γι' αυτό λοιπόν και εξαιρούνται τα χταπόδια. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να λειτουργεί η εταιρική σχέση. Ποια μορφή πρέπει να λαμβάνει η αλληλευτική πολιτική και πώς ακριβώς πρέπει να επιδιώκουμε την βιώσιμη αλεία. Για άλλη μια φορά λοιπόν ευχαριστώ την εισηγήτρια και περιμένω να δω με ενδιαφέρον την κριτική που θα ασκήσει η Επιτροπή Αλίας. Αλλά κατά τη δική μας την άποψη όλα αυτά είναι θετικά και βρισκόμαστε σε έναν όπως σας είπα καλό υποδειγματικό μάλλον δρόμο. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου Θα ήθελα να ξεκινήσω με τα συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια την κυρία Μάισναρ για το περιεχόμενο του κειμένου. Όπως αναφέρθηκε, ε, πρέπει τώρα να συζητήσουμε ένα κείμενο το οποίο έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της 26ης Ιουνίου ε, του έτους που εκπνέει. Και είναι σημαντική η συμφωνία αυτή από οικονομική άποψη με μια τρίτη χώρα. Πρόκειται, όπως όλοι γνωρίζουμε και όπως ήδη αναφέρθηκε, πρόκειται για ένα θέμα που είναι ευαίσθητο, λεπτό για κάποιες χώρες μέλη και τούτο Αποδείχθηκε και στη συζήτηση στην Επιτροπή Αλληλείας, από την οποία μόλις έρχομαι. Και πρότεινα ε, τις απόψεις των φορέων αλληλείας των ευρωπαϊκών χωρών, κάτι το οποίο ε, είχε απήχηση και στον ευρωπαϊκό τύπο. Πρέπει να πούμε ότι το Σεπτέμβριο του 2012 οι Μαυριτανοί αλληλείς οργάνωσαν μία πορεία υπέρ της υποστήριξης του πρωτοκόλου που υπογράφεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαυριτανίας. Πρόκειται δηλαδή για μία θετική κίνηση. Και επίσης οι εκπρόσωποι τους ε, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι το κείμενο αυτό ε, λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των φτωχών και προσφέρει δυνατότητες στους ε, ε, αλλιευτικούς φορείς της Μαυριτανίας και τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν. Και στις συναντήσεις που είχαμε με τους εκπροσώπους της χώρας υπό την αιγίδα των υπευθύνων φορέων για τις χώρες Μαγκρέμπ επιβεβαιώθηκε η ικανοποίηση αυτή ως προς τα σκάφη τα οποία λειτουργούν στα κινούνται και αλλιεύουν στα μαυριτανικά ύδατα. Και βεβαίως η συμφωνία αυτή είναι θετική και για την ευρωπαϊκή πλευρά. Θέλω εδώ να υπενθυμίσω τις συζητήσεις που οργανώθηκαν στην Επιτροπή Αλίας, διότι εκεί υπήρξαν τέσσερα επιχειρήματα. Τέσσερα επιχειρήματα που ουσιαστικά εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς το πρωτόκολλο αυτό. Ε, και, και ακόμα θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, ότι διατυπώθηκαν και πολύ αρνητικές απόψεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν κατάλαβα καλά, ένα πρώτο επιχείρημα είναι ότι πρόκειται για μια συμφωνία που καθιστά το πρωτόκολλο πολύ πιο ακριβό από ό,τι το προηγούμενο. Δεύτερον, δεν ε, λαμβάνονται υπόψη πολύ σοβαροί τεχνικοί περιορισμοί. Τρίτον, η ιδέα απαγόρευσης αλίευσης κεφαλοπόδων ε, δεν βοηθάει τις, τις μικρές πυρόγες που χρησιμοποιούν οι Μαυριτανοί, δηλαδή τα μικρά σκάφη, αντιθέτως ε, βοηθά τον κινέζικο στόλο. Και επίσης ένα άλλο επιχείρημα που διατυπώθηκε στην Επιτροπή Αλίας είναι η υποχρέωση, ε, η υποχρέωση το 2% των ε, πελαγικών αλλιευμάτων, το 2% λοιπόν των αλλιευμάτων να διατίθεται στην ε, μαυριτανική αγορά. Και συζητήθηκαν οι συνέπειες που μια τέτοια απόφαση μπορεί να έχει για μια μικρή χώρα όπως η Μαυριτανία. Ιδού λοιπόν αυτές ήταν οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στην Επιτροπή Αλίας. Εδώ τώρα στην Επιτροπή Ανάπτυξης ακούσαμε θετικά σχόλια και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη στις χώρες εταίρους. Και η Μαυριτανία είναι μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και ο τομέας της αλληλείας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, το 1 τέταρτο του ΑΕΠ και εξασφαλίζει ε, περίπου 36.000 θέσεις απασχόλησης. Εδώ λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και θα ήθελα να επισημάνω και ένα σημείο που η συγγήτρια κυρία Μάιστερ και η ίδια υπογράμμισε, την ανάγκη δηλαδή της συνέπειας. Καταρχήν με τον εαυτό μας η συγγήτρια ε, αναφέρθηκε στο ψήφισμα που εγκρίναμε στις 12 Μαΐου του 2011. Και επίσης ε, συνοχή με τη δική μας αναπτυξιακή πολιτική, διότι ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να, το πρωτόκολλο αυτό και το περιεχόμενό του να εμπίπτει και στις αρχές της συνθήκης. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δίδεται η έγκριση στο, για το πρωτόκολλο αυτό, το οποίο δίνει κάθε δυνατότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και οι τρεις συστάσεις που κάνει η συγγήτρια στο τέλος μου φαίνονται επίσης θετικές για να βελτιωθεί το κείμενο. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ να αγνοήσω το γεγονός ότι η Επιτροπή Αλίας βρίσκεται σε ένα άλλο πεδίο, αν θέλετε. Ε, ε, αισθάνθηκα την υποχρέωση να τα πω αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νιούτον Ντάν έχει το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ την ε, φίλη και εισηγήτρια. Μία ερώτηση. Τις προάλλες πήρα ε, μία επιστολή από έναν από την εκλογική μου περιφέρεια που κατηγορούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρησιμοποιεί την τεράστια ισχύ που έχει ε, απέναντι στην, στο Μαυρίκιο, όχι τη χώρα που αναφέρατε εσείς, τη, Μαυριτανία, και είπατε ότι, ότι έχουμε απίστευτες εξουσίες για να εκμεταλλευόμαστε τους α, καημένους ψαράδες, ας πούμε, του Μαυρίκιου. Πώς το κάνετε αυτό. Ε, του είπα δεν έχω καμία ιδέα. Ε, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι ο λαός της Μαυριτανίας είναι ικανοποιημένος με αυτή τη συμφωνία. Ναι, είναι ικανοποιημένη με αυτή τη συμφωνία. Ε, να μιλήσω γερμανικά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, όπως μου δείχνει εδώ και ο βοηθός μου, ότι υπήρξε μια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που ελήφθη υπόψη. Άρα δηλαδή εγώ στην έκθεσή μου έλαβε υπόψη μου τα συμπεράσματα. Ε, κατόπιν του εγώ θέλω να σας πω, οι Μαυριτανοί είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό και σας το είπα και πριν ότι ήταν, ε, εμφανίστηκαν στις διαπραγματεύσεις με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ξέρω ότι στην Επιτροπή Αλίας η προσέγγιση είναι διαφορετική, τα επιχειρηματά τους είναι τελείως διαφορετικά. Ξέρετε γιατί, γιατί θίγονται τα ευρωπαϊκά του συμφέροντα. Πάντως από πλευρά αναπτυξιακής για να είμαστε ε, συνεπείς ε, πρέπει να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία. Δεν πρόκειται για το Μαυρίκιο. Άλλο ο Μαυρίκιο, άλλη Μαυριτανία. Τώρα μιλάμε για τη Μαυριτανία, λέει ο Μιλίτρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ε, πρόεδρε, συγγνώμη. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο επίσης στη συζήτηση. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη θέση της Επιτροπής σας. Αυτό το πρωτόκολλο με τη Μαυριτανία είναι το πρώτο πρωτόκολλο που έχει την αηφόρη αηφόρα διάσταση μέσα του και που λαμβάνει υπόψη τις νέες ε, αρχές της εξωτερικής διάστασης της ε, πολιτικής αλίας, κυρίως τα πλεονάσματα, ότι η τρίτη χώρα θα πρέπει ε, να λάβει υπόψη τις δικές της ανάγκες και να εκφράζονται αυτές στις συμφωνίες και όλα τα θέματα που συνδέονται με την περιβαλλοντική προστασία. Είμαι ικανοποιημένη λοιπόν που συμμερίζεστε αυτή την άποψη μαζί μας. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποιες μικρές ε, διευκρινήσεις σε σχέση με αυτά που είπε η συγγητριά σας. Καταρχάς, κυρία Μάιστερ, μιλήσατε για τη μεταβατική περίοδο, η οποία παρατείνεται μέχρι το τέλος ε, του Ιανουαρίου. Άρα πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Να πω σε όλους σας εδώ ότι το πρώτο κόλλο με τη Μαυριτανία υπογράφτηκε χθες. Ε, στη Μαυριτανία η Κυριακή είναι εργάσιμη ημέρα και το υπογράψαμε χθε λοιπόν στη Μαυριτανία. Από σήμερα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε τις αλληλευτικές μας δραστηριότητε. Αυτή η μεταβατική περίοδος λοιπόν τέλειωσε. Δεν υπάρχει. Και το πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ. Υιοθετήθηκε προσωρινά από το Συμβούλιο και υπογράφτηκε. Τώρα λοιπόν το μπαλάκι είναι στο κοινοβούλιο, το οποίο θα πρέπει να δώσει τη συνένεσή του ή όχι. Ελπίζω λοιπόν μαζί να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να δώσει θετική γνώμη το Κοινοβούλιο για αυτό το πρωτόκολλο. Δεύτερον, θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην ε, στήριξη του κλάδου. Τα χρήματα δηλαδή που ξεπερνούν τα εμπορικά θέματα και που δίδονται για την ανάπτυξη του κλάδου της αλίας. Η κυρία Μάισνερ πολύ σωστά είπε ότι αυτός ο τομέας, αυτή η πτυχή, ε, πρικοδοτείται με 3 εκατομμύρια ευρώ και εδώ έχουμε μείωση σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο που κατά μέσο όρο κατέτος δίναμε 16 εκατομμύρια. Είμαστε στην Επιτροπή Ανάπτυξης θέλω να σταθώ λιγάκι σε αυτή τη μείωση. Πώς δικαιολογείται. Υπάρχει ένας και μόνο λόγος. Η Μαυριτανία δεν χρησιμοποίησε σωστά τα 16 εκατομμύρια ετησίως που προέβλεπε το προηγούμενο πρωτόκολλο. Καταλάβαμε ότι η αλία ως κλάδος δεν ήταν η απόλυτη προτεραιότητα της Μαυριτανίας. η Μαυριτανία έχει άλλα πιο επίγοντα προβλήματα. Το σύστημα υγείας της, το σύστημα παιδείας, το σύστημα υποδομών της. Και όταν μιλάμε για το ότι η ίδια η χώρα θα πρέπει να διαχειρίζει μεγάλες, ε, τα, μεγάλα κονδύλια για την ανάπτυξη, σε αυτό το πλαίσιο η Αλία έχει μόνο έχει δεύτερη θέση. Αυτό το κατέδειξε σαφώς το προηγούμενο πρωτόκολλο, γι' αυτό μειώσαμε το ποσό που δίνουμε στην ε, τομιακή στήριξη. Δεν υπήρξε αυτή η μείωση γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη. Όχι, υπάρχουν ανάγκε. Απλώ η Μαυριτανία θεωρεί ότι αλλού είναι οι προτεραιότητε. Ένα πολύ λεπτό θέμα είναι τα κεφαλόποδα. Η Μαυριτανία μα είπε ξεκάθαρα ότι σκοπεύει να αναπτύξει τον τομέα της ε, τεχνικής αλίας. Δηλαδή θέλει να δώσει προτεραιότητα στους ντόπιου ε, ψαράδες για να ψαρεύουν τα κεφαλόποδα. Αυτοί οι αλεί έχουν την ικανότητα να ψαρεύουν το σύνολο των κεφαλόποδων. Άρα τι να πούμε. Έχουν κάθε δικαίωμα. Το καθήκον μας είναι να τους υποστηρίξουμε. Σε ό,τι αφορά την ε, τον κλασικό ε, αλλιευτικό στόλο ε, που είναι κινέζικης προέλευσης. Γιατί το λέμε εδώ μεταξύ μας, ε, εν πάση ειλικρινία, ότι η Μαυριτανία δεν, είναι, δεν έχει δικό της στόλο που μπορεί να τον οικοδομήσει με δικά της κονδύλια, με δικά της χρήματα, αλλά οι Κινέζοι φτιάχνουν αυτά τα πλοία και τα πλοία αυτά φέρουν τη σημαία της Μαυριτανίας. Έτσι. Η Μαυριτανία αυτή τη στιγμή ξεφορτώνεται τα παλιά κινέζικα ε, σκάφη, τα οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση και τα οποία δεν σέβονται τις, ε, τους κανόνες υγιεινής που επιβάλλει η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Αυτά τα πλοία θα εξαφανιστούν, θα παροπλιστούν και ίσως υπάρξουν νέα σκάφη. Μάλλον θα ξέρετε ότι θα υπάρξει μια νέα σύμβαση με την Κίνα, η οποία θα υπογραφεί, αλλά προς το, προς το παρόν πρέπει να σας πω ότι η Μαυριτανία μείωσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Κίνα. Προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει αν ε, θα οικοδομηθούν νέα κινέζικα σκάφη για να ψαρεύουν τα κεφαλόποδα. Εμείς θα ενθαρρύνουμε τη Μαυριτανία ούτως ώστε να δώσει προτεραιότητα στην ε, ανάπτυξη α, της μικρής ερασιτεχνικής που ψαρεύει κεφαλόποδα εις βάρος της βιομηχανικής, ας πούμε, εντατικής αλίας. Αν ληφθεί από τη Μαυριτανία πολιτική απόφαση να αναπτύξει παράλληλα με τα μικρά σκάφη και μεγάλα σκάφη, με τη σημαία της, που τα φτιάχνουν άλλοι, ε, εμείς τι να κάνουμε, πρέπει να σεβαστούμε αυτή την επιλογή της τρίτης χώρας. Τώρα, τα δύο-τρία σημεία που ανέφερε ο κύριο Φρέντα. Ξέρω ότι εδώ δεν είσαστε η Επιτροπή Αλία, αλλά θέλω να σχολιάσω κάποια από αυτά που είπατε. Το πρωτόκολλο δεν κοστίζει πιο ακριβά. Αντικατοπτρίζει απλώ καλύτερα την πραγματική τιμή του ψαριού. Και δεν είναι σωστό ότι όλες οι αλλιευτικέ ευκαιρίε εξαφανίζονται. Υπάρχουν, ας πούμε, περισσότερα πελαγικά ε, ψάρια. Απλώς γίνεται μια αναδιάρθρωση, μια προσαρμογή. Μπορεί οι τεχνικέ προδιαγραφέ να φαίνονται πιο επαχθεί ε, για τον κλάδο, αλλά το κάνουμε αυτό για λόγου αηφορία. Αυτή είναι η δικαιολογία. Η Κομισιόν θα πρέπει να προτάξει τους, ε, τα εμπορικά, ας πούμε, συμφέροντα του στόλου, που θα κατασπαράξουν, ας πούμε, και τους πόρους ε, και τα νερά ή θα πρέπει να προωθήσουμε την αηφόρο προσέγγιση. Το 2% των ψαριών που θα τα δίδουμε στη Μαυριτανία. Δεν πάνε στην αγορά. Θα τα μοιράζουμε δωρεάν στον πληθυσμό. Θα υπάρξει ένα σύστημα διανομής ψαριών δωρεάν στον πληθυσμό που έχει ανάγκη. Αυτά τα λιεύματα λοιπόν δεν θα δημιουργήσουμε ανισορροπία στην αγορά τη Μαυριτανία. Αυτά σα ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σα αν έχετε και άλλε ερωτήσει. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να κάνω μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Δηλαδή, Πώς μπορούμε εμείς ε, να επηρεάσουμε αυτή τη ε, συμφωνία μεταξύ Μαυριτανίας και Ευρωπαϊκού Στόλου. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ενδεχομένω να προκύψουν και θέματα απασχόλησης. Κατόπιν, όσον αφορά την υπεραλήψη των ε, κεφαλόποδων στην περιοχή, αυτό αποτελεί Υπάρχει κίνδυνος για αυτό το είδος ψαριών ή όχι. Κινδυνεύουν αυτά τα ψάρια ή όχι. Και κατόπιν, αυτά τα 2% ε, που διανέμονται στους ε, πολίτες της ε, Μαυριτανίας. Εκεί μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά κάποια λύση για να αλλάξει την τιμή και αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο η Κομισιόν μήπως τελικά δημιουργήσει και πρόβλημα στη Μαυριτανία. Πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή να απαντήσει, παίρνω το λόγο εγώ. Θυμάμαι ότι κατά τη διάρκεια ε, της δικής μου θητείας είχα τη συμφωνία αλλιές με την ε, Λοιπόν, και πρέπει να πω ότι η συμφωνία με τη Μαυριτανία και το κείμενο της συναδέλφου κυρία Μάισνερ είναι ένα ισορροπημένο κείμενο που λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και τους πόρους και την βιωσιμότητα και αυτό είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγητριά μας για τη σύνταξη της έκθεσης δεδομένου ότι έλαβε υπόψη τις ε, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις και αυτό είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό, να βλέπουμε δηλαδή τις διαστάσεις αυτές να περιλαμβάνονται σε μια αλλιευτική συμφωνία. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για αυτά τα πολύ ενθαρρυντικά σχόλια, τα, παρα... τα... τα αναμένουμε πάντοτε με ευχαρίστηση. Απαντώντας τώρα στις ερωτήσεις. Ναι, πράγματι θα υπάρχει μια επίπτωση στα σκάφη. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τα κεφαλόποδα είναι συγκεκριμένα και το πρωτόκολλο καθώς εξέπνε στις 31 Ιουλίου ε, δεν υπήρχε δυνατότητα αλληλείας ε, κεφαλόποδων και για ένα αρκετά βέβαιο μέλλον. Ε, και εάν συνεχιζόταν αυτό, η Μαυριτανία ως κυρίαρχο κράτος μπορούσε να λάβει ε, αποφάσεις, κυρίαρχες αποφάσεις. Δεν βρισκόμαστε στην απεικιοκρατική περίοδο και δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε στη Μαυριτανία το τι ακριβώς θα πράξει. Τώρα, ως προς την ε, ε, χρηστή διαχείριση των ε, θεμάτων κεφαλοπόδων στην ε, Μαυριτανία. Εμείς ε, καταγράφουμε στο πρωτόκολλο πώς δηλαδή η Μαυριτανία θα εκμεταλλευτεί τα, ε, τους καρπούς της αλίας με βιώσιμη εκμετάλλευση κάθε είδους περιλαμβανομένης και της αλίας των κεφαλοπόδων. Τώρα, ως προς το 2% της δωρεάς τούτο δεν αφορά στα κεφαλόποδα. Και είναι λογικό, διότι δεν αλλιεύονται πλέον αυτά. Μόνον, αφορά μόνο στα μικρά πελαγικά ψάρια. Τα μικρά ψάρια τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια και που δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία και που αυτά διανέμονται στην Μαυριτανία. Και δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, διότι οι Μαυριτανοί είναι νομάδες της ερήμου ε, φοβούνται τη θάλασσα, δεν την εκμεταλλεύονται και δεν τρώνε και πολλά ψάρια. Συνεπώς η αγορά ψαριών της Μαυριτανίας δεν υφίσταται ουσιαστικά και επειδή αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η χώρα μια οξία ε, κρίση τροφίμων, αυτή η κίνηση διάθεση του 2% και απαντώ στον κύριο Πρέντα, εξηγώ δηλαδή και εκφράζω την ίδια άποψη, αυτή η δωρεά λοιπόν του 2% δεν πρόκειται να διαταράξει την αγορά ηχθείων της Μαυριτανίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάισνερ, τώρα έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εγώ είχα επισημάνει τις ε, δυσκολίες ε, που θα προέβαλαν ε, και που υπάρχουν πράγματι από σκοπιά. Σας το είπα πριν, άλλο ελεκτική, άλλο ενεπτυξιακή σκοπιά. Κοιτάξτε, εμείς ως Κοινοβούλιο μπορούμε να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Προφανώς ε, θα ήταν καλύτερα κι εσείς ε, να περιμένατε να ακούσετε και την άποψη του Κοινοβουλίου. Ε, αυτό είναι πολύ γενικό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας είπα, για τους λόγους που σας εξήγησα, είναι καλύτερα από αναπτυξιακή σκοπιά να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει μία προθεσμία μέχρι 9 Ιανουαρίου ε, το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 18 Φεβρουαρίου. Και περνούμε τώρα στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης. Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική είναι το θέμα. Η συγγήτρια στο θέμα αυτό είναι η κυρία, κυρία Κορίνα Κρετού. Δεν είναι σήμερα παρούσα. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα την αντικαθιστά. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Γυναικών που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Ο κύριος Κόρτες Λάστρας έχει το λόγο αμέσως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όπως είπατε κι εσείς, η κυρία Κρέτου είναι η συγγήτρια για την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι παρούσα, όπως είπατε, και μου ζήτησε να σας ζητήσω συγγνώμη για την απουσία της στην ε, συζήτηση. Λοιπόν, τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά σήμερα που ζούμε σε οικονομική, χρηματοπιστωτική και ανθρωπιστική κρίση. Η πλήρης ε, χρήση των εργατικών χεριών των γυναικών είναι σημαντικό για την εξάλληψη της στόχιας και την αύξηση του ανταγωνισμού και μάλιστα ενός βιώσιμου ανταγωνισμού. Στη Βόρεια Αφρική ε, αυτή είναι μια περιοχή όπου τίθενται πολλά προβλήματα ισότητας φύλων. Ευτυχώς όμως υπάρχουν α, ε, οργανώσεις και μετά την Αραβική Άνοιξη ε, τίθενται αυτά τα θέματα για την ε, πολιτική και νομική προστασία των γυναικών. Κάθε μέρα βλέπουμε ε, ποια είναι τα δύναμα, ότι οι γυναίκες είναι αδύνατες στις χώρες αυτές. Στην Αίγυπτο, ας πούμε, ε, δεν υπήρχε καμία γυναίκα στην Επιτροπή η οποία ε, εκπώνησε την, το σχέδιο συντάγματος. Ε, βέβαια, η κατάσταση από χώρα σε χώρα διαφέρει. Ε, η συμμετοχή όμως των γυναικών στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων υπόκειται σε διάφορες προϋποθέσεις για να επωφεληθούμε από το δυναμικό που έχουν οι γυναίκες. Η Κορίνα λέει ότι καταρχάς θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι τα κοριτσάκια πηγαίνουν στο σχολείο ε, με κατάλληλα εργαλεία και προγράμματα και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ε, καλά μοντέλα, καλά πρότυπα τα οποία περνάνε μέσα από τα σχολεία για τις γυναίκες. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα ενημερωτικά, θα πρέπει οι γυναίκες δηλαδή να, είναι, να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες. Θα πρέπει επίσης να έχουν ίση πρόσβαση στο, στις ιατρικές υπηρεσίες, στην δικαιοσύνη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, η Κορίνα λέει ότι υπάρχει ένα κενό σε ό,τι αφορά την, τα δικαιώματα των γυναικών στην νομοθεσία. Ε, σχεδόν δεν υπάρχουν πουθενά, δεν έχουν θέση ούτε στην πολιτική ζωή, ούτε κατά την εκπόνηση των νόμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει βιώσιμα μέτρα, ούτως ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό και να ε, καταπολεμήσουμε την άνηση αμοιβή, αμοιβή ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν ίση πρόσβαση στην αγορά εργασια θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και ενίσχυση της ε, κοινωνικής προστασίας. Η Κορίνα επίσης επιμένει το Κοινοβούλιο να ζητήσει από το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρξουν εθνικά ε, προγράμματα για συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών των χωρών της ε, Βορείου Αφρικής. Είναι σημαντικό αυτό για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι θετικό το ότι ε, βελτιώνονται οι στρατηγικές της Κομισιόν, τόσο ώστε να υπάρχουν εθνικά προγράμματα εργασίας και την ε, συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών. Επίσης, η συγγήτρια θα παρουσιάσει μια τροπολογία, ούτως ώστε να εξειδικεύσει και να προσδιορίσει την παράγραφο 7. Κυρία Πρόεδρε, θα μας πείτε και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για τροπολογίες κτλ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαμπρόφσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι οι θέσεις αυτές είναι πολύ ισορροπημένες και πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση περιλαμβάνει πράγματα που λείπουν από την έκθεση. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Γυναικών και τα σημεία που ανέφερε η κυρία Κρέτσου στην γνωμοδότηση της δικής μας Επιτροπής είναι ακριβώς αυτά που έλειπαν στη θέση που παρουσίασε η κυρία Κώστα. Η αρχική έκθεση είναι πολύ πολιτικοποιημένη και απεικονίζει την κατάσταση στην ε, Βόρεια Αφρική, ε, όπως διαμορφώθηκε τον τελευταίο χρόνο. Ξέρουμε όμως ότι τα προβλήματα των γυναικών είναι πολύ βαθύτερα, πολύ παλιότερα, δεν είναι μόνο της τελευταίας χρονιάς φυσικά. Και επηρεάζονται πολύ από την ε, κουλτούρα της περιοχής. Εγώ ξέρω αυτή την περιοχή γιατί δούλεψα ως γιατρός επί τέσσερα χρόνια στη Βορειοαφρική. Και τα προβλήματα που αναφέρει η κυρία Κρέτσου είναι πραγματικά τα πιο σημαντικά. Ίσως στο σημείο 5 θα έβαζα μεγαλύτερη ε, έμφαση στις μικροπιστώσεις. Αναφέρει τα προγράμματα που εστιάζουν στην ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αλλά νομίζω ότι το θέμα των μικροπιστώσεων και μικροδανείων είναι πολύ, πιο... είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να του δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Είναι σημαντικό όχι μόνο για να εκπαιδευτούν και να καταπιστούν οι γυναίκε, αλλά του δίνει και κάποια αρχικά ας πούμε, κονδύλια για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Μπορώ να το υποβάλω αυτό ως μια τροπολογία στο κείμενο της κυρίας Κρέτσου. Πιστεύω πάντως ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι ένα πολύ καλοδιατυπωμένο κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Η κυρία Ραφαέλα Ιώδης. Yes, Ευχαριστώ. Ακούσαμε την έκθεση και συμμεριζόμαστε πλήρως τις απόψεις της εισηγήτριας. Η Επιτροπή αυξάνει τη στήριξή της προς τις γυναίκες. Φυσικά το θέμα αυτό είναι οριζόντιο εν υπάρχει σε όλα τα προγράμματα και πάντα σε όλα τα προγράμματα μας υπάρχει η διάσταση του φύλου. Ε, εγώ γνωρίζω την περιοχή, ήμουν εκεί τα τελευταία εννέα χρόνια, μόλις επέστρεψα και γνωρίζοντάς την μπορώ να πω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Την λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την έκθεση πάντως. Θα ήθελα μέσα σε ένα λεπτό να υπενθυμίσω ότι έχουμε 92 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα περιφερειακής και διμερής ε, συνεργασίας. Πριν από ένα μήνα ε, δώσαμε μία επιχορήγηση για να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή και να βελτιώσουμε τα δικαιώματά τους ε, στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος του ΟΗΕ. Αυτό. για όλες τις γυναίκες στην περιοχή αυτή, όχι μόνο στις πρωτεύουσες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα για να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Όχι. Υπεν... Όχι. Υπενθυμίζω ότι έχετε μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 10 η ώρα ε, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών και η έκθεση θα ψηφιστεί στις 22 Ιανουαρίου. Και ερχόμαστε τώρα στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης σχετικά με την πλατφόρμα για την εξωτερική συνεργασία και την ανάπτυξη. Μετά από το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την πλατφόρμα για την εξωτερική συνεργασία και την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Οκτωβρίου μια επιτροπή, ε, συγγνώμη, επιστολή που περιέχει ακριβώς το περιεχόμενο αυτής της πλατφόρμας και τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας. Η επιστολή αναφέρεται στους ε, επίσημους μηχανισμούς και η ανταλλαγή απόψεων τώρα θα βοηθήσει ε, στο να δώσουμε περιεχόμενο σε αυτή την πλατφόρμα. Ο κύριος Στάση ήταν ε, ο εισηγητή από πλευρά της Επιτροπής μας και επειδή σήμερα δεν είναι παρόν μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Ο κύριος ε, Ζέμ Κόντε, επικεφαλής της ε, μονάδας για τα χρηματοοικονομικά μέσα στην ε, EuroPaid, θα μας παρουσιάσει τους στόχους και τους τρόπους λειτουργίας αυτής της πλατφόρμας, η οποία EuroPaid συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 14 Δεκεμβρίου. Ε, στη συνέχεια θα λάβει το λόγο ο κύριος Αλασάνδρο Καράνο, επικεφαλής της μονάδας της, ε, της, επικεφαλής της ε, διεύθυνσης για τις πολιτικές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα θεσμικά θέματα και μετά η κυρία Κατρίν Κολέν, επικεφαλής του Τμήματος Συντονισμού ε, των δραστηριοτήτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το, χρόνο, το λόγο για 10 λεπτά. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο θα αναφερθώ αμέσως στους στόχους της πλατφόρμας έτσι όπως τις ε, συλλάβαμε και καθορίστηκαν στο πλαίσιο της εργασίας, της ομάδας εργασίας ε, που δούλεψε μεταξύ Νοεμβρίου και Ιουνίου. Βασικό στόχος είναι να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ε, μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτικό πλαίσιο που καλύπτει τις σχέσεις με τις χώρες εταίρους. Έτσι λοιπόν, καλύπτει η πλατφόρμα βάσει ε, της απόφασης της ε, Κομισιόν ε, δραστηριότητες γειτονίας με τις χώρες εταίρους. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα θα καλύπτει όλες τις περιοχές εκτός Ευρώπης, εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται στην ανάπτυξη ε, και έχει αναπτύξει σχέσεις με τις γειτονικέ χώρες. Έτσι λοιπόν, καλύπτει όλους τους τομείς που, έχουν, που επηρεάζουν την ανάπτυξη και συνδυάζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Στόχος είναι να βελτιωθεί η απόδοση των υπαρχόντων μέσων χρηματοδότησης, η εναρμόνιση τους με τις, η αρμονική μάλλον ανάπτυξή τους με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Η πλατφόρμα θα καλύπτει τι ε, δικαιούχους χώρες. Στο πλαίσιο αυτής της ε, προσπάθειας ανάπτυξης, όπως λέει, ε, ανάμιξης, blending ή mixage. Ε, θα γίνει χρήση λοιπόν των υπαρχόντων μηχανισμών και εκεί όπου χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις, Σύμφωνα με τις συστάσεις της πλατφόρμας θα γίνεται προσφυγή στις υπάρχουσες δομές, είτε δηλαδή στις Επιτροπές Διαχείρισης, είτε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη σκοπιά της δομής συγκροτήθηκε μια ομάδα εργασίας που χωρίστηκε στα δύο. Μια ομάδα πολιτικής, στην οποία συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες μέλη, και υπάρχει και ένας παρατηρητής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την άλλη υπάρχει τεχνική ομάδα που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στα διάφορα επενδυτικά προγράμματα. Η γραμματεία των δύο αυτών υποομάδων θα καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, όπως ήδη αναφέρθηκε από την κυρία Πρόοδο, η πρώτη συνεδρίαση της πλατφόρμας έλαβε χώρα την Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας, 14 Δεκεμβρίου, με την ε, συγκρότηση έγινε και μια πρώτη συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας. Μετά παρουσιάσαμε την τα διάφορα μέσα χρηματοδότησης στις διάφορες περιοχές, υιοθετήσαμε ένα πλάνο εργασίας, όχι επίσημα, διότι αυτά όλα πρέπει να γίνουν ε, γραπτά, αλλά υπάρχει ευρεία συμφωνία και συνένεση για το πρόγραμμα εργασίας του 2013. Και έτσι λοιπόν με τη συγκρότηση των δύο υποομάδων που σας ανέφερα, η μία ομάδα θα εξετάσει τους μηχανισμούς blending, ανάμιξης, μιξάζ, αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων ως προς την απόδοσή τους, θα εντοπίσει βέλτιστες πρακτικές και επίσης άλλες πτυχές οι οποίες δεν αποδίδουν ικανοποιητικά μέχρι τώρα. Ενώ η δεύτερη ομάδα σχετικά με την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων ανάμιξης, blending, mixage, ε, αυτή η δεύτερη ομάδα θα εφαρμόσει ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων με τυποποιημένο τρόπο. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει συνεργασία με τα χρηματοοικονομικούς φορείς και ήδη θα υπάρχει μια συνάντηση τον Ιανουάριο. Η πρώτη ομάδα θα εξετάσει τους υπάρχοντες μηχανισμούς blending και θα εκεί θα προεδρεύει η Κομισιόν, ενώ η Κομισιόν έχει την πρόθεση να προτείνει το προεδρείο αυτής της ε, ομάδας να είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Καράνο και την κυρία Κολάν, τους οποίους παρακαλώ να μοιραστούν το χρόνο των 10 λεπτών. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ που μας ε, καλέσατε και ε, μας δώνετε τη δυνατότητα να έρθω στην Επιτροπή ε, την Αναπτυξιακή σχετικά με το μείγμα αυτό ε, ανάμεσα στις ε, δόσεις και τα δάνεια που χορηγούνται. Όπως ξέρετε, εμείς έχουμε ένα πλαίσιο για δανειοδοτήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως αυτές που αφορούν την εξωτερική εντολή. Αυτό προβλέπεται ε, σε σχέση με τη διεύρυνση και τις ε, γειτονιάσεις ε, περιοχές προβλέπεται η Συμφωνία ΑΚΕ και σε σχέση με τη Συμφωνία Κοτονίου. Εμείς λοιπόν χορηγούμε δάνεια σε συνδυασμό με κονδύλια του προϋπολογισμού και αυτό για να στηρίξουμε τις βιώσιμες επενδύσεις. Αυτό το κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό και εστιάζουμε την προσοχή μας κυρίως σε τρεις τομείς. Ο ένας είναι η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα που όπως πολύ καλά γνωρίζετε συμβαδίζει και με το νέο θεματολόγιο για, τον, ε, για την αλλαγή του προσανατολισμού. Μας ενδιαφέρει επίσης η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής και η υποστήριξη των επενδύσεων ε, στην κλιματική προσαρμογή και την άμπλυνση των κλιματικών επιπτώσεων. Η συνάδελφός μου θα αναφερθεί στα θέματα της χρηματοδότησης. Τώρα όσον αφορά τις δραστηριότητες μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάμε για ένα ποσό των 8 δις ε, σε αιτήσια βάση. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα τρίτο των δραστηριοτήτων της Παγκόσμιας Τράπεζας κατά μέσο όρο τα τελευταία πέντε έτη. Αν προσθεθούν και δικέ μας οι δραστηριότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα ε, Ανασυγκρότησης mainly Uh, Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναπτύσσει μια μεγάλη δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν συμμετέχουμε από το 2007 σε διάφορα εργαλεία μίξης ε, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αφρική, για τις γειτονικέ περιοχές, για τα Δυτικά Βαλκάνια και για άλλες ε, περιοχές. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι αυτά όλα πολύ σημαντικά έτσι ώστε να υπάρξει μόχλευση της οικονομικής δυνατότητας και της Εμπειρογνωμοσύνης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αυτά σε συνδυασμό ε, με άλλες ε, τραπεζικές δραστηριότητες. Εμείς ε, θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση έτσι ώστε να συσχετίζονται οι πολιτικές προτεραιότητες και ο προσανατολισμός μέσα από πρακτική χρηματοδότηση επενδύσεων. Εξάλλου, Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους χρηματοπιστωτικούς ε, θεσμούς και οργανισμούς, καταρχήν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό είναι απόλυτα σαφές, αλλά και με άλλα Ινστιτούτα ιδιωτικά, αλλά και δημόσιου χαρακτήρα. Βεβαίως, εξακολουθούμε να έχουμε διαφορετική προσέγγιση εμείς σε σχέση ε, με άλλους οργανισμούς όσον αφορά την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εμείς, όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα, αυτό θα πρέπει να προβάλλεται ε, στις ε, χώρες μέλη όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. Άρα, δηλαδή, λειτουργούμε συντονισμένα. Σας είπα για να υπάρξει μόχλευση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των οικονομικών πόρων που είναι απαραίτητη ε, η μόχλευση και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα καθίστανται όλο και σημαντικότερα στοιχεία. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει και είμαστε και δεσμευμένοι είναι να εφαρμόζουμε τις ε, πολιτικές και τις προδιαγραφές ανάλογα με αυτά που μας λένε οι μέτοχοί μας και δεσμευόμεθα από ελέγχους ε, που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από το Διαμεσολαβητή και άλλους. Επιπλέον, εμείς ε, έχουμε πρόσβαση σε πιστώσεις μόνο εφόσον εγκρίνονται από τον κοινοτικό προπολογισμό ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ άλλοι θεσμοί έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια των μετόχων. Θέλω να υπογραμμίσω, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε ε, να αλληλοσυμπληρωνόμαστε μετά για, την εκτέλεση των ίδιων προγραμμάτων, γιατί περίπου το 40% των δικών μας προγραμμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδοτούνται και από άλλους ε, θεσμούς. Άρα υπάρχει περιθώριο συγχρηματοδότησης. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δικές μας τράπεζες και τους άλλους θεσμούς. Ε, στο επόμενο σε δημοσιονομικό πλαίσιο ελπίζουμε να υπάρξει μια μεγαλύτερη ανάμειξη όλων αυτών των δυνατοτήτων και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει τις εξωτερικές δραστηριότητες 14 20 που θα συζητηθούν την επόμενη χρονιά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μας στηρίξετε και η συνάδελφός μου θα συνεχίσει με συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα. Ευχαριστώ Αλεσάνδρο, σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την ε, Κομισιόν ε, χρονολογείται ε, από πολύ παλιά. Ε, του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 50 χρόνια ε, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τις χώρες ΑΚΕ. Αυτή η συμφωνία συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ΑΚΕ. Ε, είναι η πιο παλιά συμφωνία, στο μεταξύ όμως, μετά όμως υπήρξαν και άλλες συμφωνίες. επίσης, Ένα άλλο από τα εργαλεία ανάμειξης, blending, που δημιουργήθηκε είναι το καταπίστευμα για τη τις επενδύσεις στην Αφρική. Υπάρχει ένα project στα πλαίσια του που χρηματοδοτείται από αυτό το καταπίστευμα και που δείχνει ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο ως ε, χρηματοπιστωτικός οργανισμός μπορούμε να υπηρετήσουμε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει προγράμματα. Είναι ένα πρόγραμμα ε, που αφορεί τις χώρες των, αφορά τις χώρες των μεγάλων λιμνών στην Αφρική για την παραγωγή υδρο, υδροηλεκτρικής ενέργειας στα σύνορα του Κονγκό και της Ρουάντας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τρεις χώρες, ε, το Κονγκό, τη Ρουάντα και τον Μπουρούντι. Είναι ένα πρόγραμμα όπου συνεργαστήκαμε πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μέσω της αντιπροσωπείας επιτροπής που ε, υπάρχει ε, τόπου το 2008. Είναι δηλαδή μια μακρόπνοη προσπάθεια γιατί κάναμε και τεχνικές μελέτες, σε συνεχεία υπήρξαν θεσμικές μελέτες και οργανωτικές μελέτες ούτως ώστε να φτιάξουμε ένα τρίτο εργοστάσιο σε αυτό το ποτάμι, το συνοριακό. πριν από πολλά χρόνια είχε φτιαχτεί το πρώτο εργοστάσιο εκεί και σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν ε, προωθήσαμε αυτά τα προγράμματα και τα έργα και συνεχεία ε, βρήκαμε και άλλους χρηματοδότες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετείχαν ε, Ευρωπαίοι, ας πούμε, την Παγκόσμια Τράπεζα, την, Ευρωπαϊ... την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, την Νοτιοαφρικανική Τράπεζα για την Ανάπτυξη και φτάσαμε σε ένα στάδιο όπου Πιστεύουμε πια ότι τα επόμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2018 ας πούμε, το εργοστάσιο αυτό υδροηλεκτρικής ενέργειας θα μπορέσει να τροφοδοτήσει την ε, περιοχή με ηλεκτρικό ρεύμα, ε, που είναι πολύ σημαντικό για μια τέτοια περιοχή. Το σημαντικό σε αυτό το έργο είναι ότι πρόκειται για ένα έργο όπου τρία κράτη κάτσα στο ίδιο τραπέζι, που δεν ε, ήταν σε πολύ καλές σχέσεις, έτσι, δεν συνεργάζονταν καλά. Τρεις υπουργοί από τις τρεις αυτές χώρες το να βρεθούν γύρω από ένα τραπέζι ήταν πολύ σημαντικό. Ε, το, όλα αυτά υπό την εποπτεία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα έργο μεταξύ πολλών άλλων που προωθούμε. Αλλά επειδή ακριβώς δεν έχω πολύ χρόνο, θα περιοριστώ μόνο στο παράδειγμα αυτό. Δεν θα σας μιλήσω για άλλα έργα και προγράμματα που προωθούμε. Ευχαριστώ. Τώρα, ας ε, εκφράσω τις απόψεις του κυρίου Πάστας. Η Επιτροπή μας χαίρεται που αυτή η πλατφόρμα ξεκίνησε τη δουλειά της με την πρώτη συνεδρίαση στις 14 Δεκεμβρίου την περασμένη εβδομάδα. Ε, ο συνάδελφος αυτός ήταν ε, παρατηρητής, είχε διοριστεί παρατηρητής σε αυτήν την πλατφόρμα, αλλά ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να παραστεί ως παρατηρητής αυτή τη συνεδρίαση. Όμως, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε την έκθεση για την πλατφόρμα μορφή επιστολής που την απίφθινε στο Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Οκτωβρίου. Αυτό δεν επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να δώσει την άποψή του με βάση την επίσημη διαδικασία, δηλαδή έκθεση και ψήφισμα στην Ολομέλεια. Το Κοινοβούλιο δεν θέλει όμως να μπλοκάρει την εκκίνηση της πλατφόρμας και γι' αυτό επιμένει από τώρα να υπάρχει μια κατάλληλη διαβούλευση ε, τα επόμενα δύο χρόνια. Κάποια κράτη-μέλη τόνισαν σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση της πλατφόρμας ότι οι προτάσεις που έγιναν από την Επιτροπή για την πλατφόρμα ε, διαφέρουν ουσιαστικά από τις συμφωνίες όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη είχαν φτάσει όταν είχαν συζητήσει στην αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου. Επομέ... Ε, επιβεβαιώνεται ότι αυτή η πρόταση της Κομισιόν είναι μια ανοιχτή βάση για διαπραγμάτευση θέλω να θέσω τα επίσημια ως πρόταση της ΔΕΒΕ για αυτή τη συζήτηση. Το όνομα το οποίο συμφωνήθηκε από τους συμμετέχοντες στην πλατφόρμα είναι πλατφόρμα για την ε, ανάμειξη των δωρεών και των δανείων στην εξωτερική συνεργασία. Η ΔΕΒΕ πιστεύει ότι αυτό το όνομα είναι πιο περιοριστικό από αυτό που είχε προβλεφθεί αρχικά και θα πρέπει να αναφέρει ρητά τον όρο ανάπτυξη μια και αφορά την, το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας και όχι άλλα μέσα που χρηματοδοτεί ο, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα για την ε, εξωτερική βοήθεια. Αυτή η πρώτη συνεδρίαση ε, εξέτασε τους διαδικαστικούς κανόνες με τους οποίους θα λειτουργεί η πλατφόρμα. Είπαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πιστεύουμε και εμείς όπως κάποια κράτη-μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είναι επίσημος φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δεσμεύεται από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και που υπόκειται και λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην πολιτική ομάδα της πλατφόρμας και θα πρέπει, όπως είπαν κάποια κράτη-μέλη στη συνεδρίαση, να ξαναδούμε αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα δεν έχει κλείσει. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό το σημείο και να αναφέρουμε τις προτεραιότητες της ΔΕΒΕ τα πλαίσια των εργασιών της πλατφόρμας για τη βοήθεια που δίνει ε, με δωρές και δάνεια. Αυτές οι προτεραιότητες είχαν αναφερθεί και στο παρελθόν σε συνεδριάσεις της ΔΕΒΕ. Πρέπει να κάνουμε όμως τώρα μια προκαταρτική ανάλυση επιπτώσεων. Θα πρέπει να υπάρχει μια συγκέντρωση των δραστηριοτήτων και να υπάρχει πραγματική, πραγματικό αντίκτυπο στην μείωση της στόχιας. Ε, η οποία θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη οικονομικών ε, και κοινωνικών υποδομών. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε στη συζήτηση με πιο λεπτομερείς προτάσεις. Υπάρχουν ε, άλλοι βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Εάν δεν υπάρχει κάποιος βουλευτής που θέλει να πάρει το λόγο, θα ξαναδώσω το λόγο στους τρεις εκπροσώπους της πλατφόρμας για τα τελευταία τους σχόλια. Αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις συμπληρωματικές, σας ακούμε. Oui, madame. je, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τα συμπεράσματά σας. Από τη σκοπιά της Κομισιόν η πιο σημαντική πτυχή είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Εδώ και ένα χρόνο κάναμε τις προκαταρτικές ενέργειες ώστε να συγκροτηθεί η πλατφόρμα. Ίσως όπως και εσείς είπατε, ίσως δεν έχουν ακόμα όλα τελειώσει και δεν είναι όλα τέλεια αλλά από τη σκοπιά της Κομισιόν και εν της προσεχικούς περίοδου δημοσιονομικών προοπτικών, θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να ξεκινήσουν οι τεχνικές εργασίες, ώστε να αναλυθούν τα υπάρχοντα μέσα και να ε, τεθεί το πλαίσιο αυτής της ε, τεχνικής ε, της ανάμιξης, του μιξάζ, του blending από την αρχή το 2014. Αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα για μας. Ε, καταγράφω και σημειώνω τα σχόλια που κάνατε και θα τα μεταφέρω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κοιτάξτε, εμείς υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την άποψη ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. Και είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι ότι οι φιλοδοξίες της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι πολύ ψηλότερες από ό,τι συμβαίνει τώρα. Συμμετέχουμε λοιπόν σε μία σειρά ανταλλαγών, ε, συμπεριλαμβανομένη τη ανταλλαγή και με το Κοινοβουλίο. Αυτό ξεκίνησε βέβαια πριν από 1,5 χρόνο με την αναθεώρηση τη εξωτερική εντολή. Η συναπόφαση, δυνατότητα συναπόφασης ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στην εξωτερική εντολή, αυτό έδωσε την ιδέα να υπάρχει συμμετοχή στην πλατφόρμα. Και εμεί συμμετείχαμε ενεργά στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι θα υπάρξει μέσα στην πλατφόρμα ένας πυρήνα ενωσιακό, θεσμών συμπεριλαμβανομένη και τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα συμμετέχουν στον ορισμό του πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τους πόρους μας, ε, τις οικονομικές και τεχνικές μας δυνατότητες, όλα αυτά προς όφελος των εξωτερικών πολιτικών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια των πολιτικών αυτών. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρότασή σας. Ε, η EIB ε θα παίξει σημαντικό ρόλο και στις δύο αυτές ομάδες. Και αυτό ήταν η δική σας πρόταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους προσδίδω ιδιαίτερη σημασία στην πλατφόρμα αυτή. Οκτώ δις που μπορούμε να επενδύσουμε και να τα αναμίξουμε με τις δωρεές μας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να κατέχει μια ιδιαίτερη θέση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να ε, συνδυαστεί με τα άλλα χρηματοδοτήματα. Ε, χρηματοοικονομικά όργανα για να έχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν θα διακόψουμε την συνεδρίασή μας και θα επαναλάβουμε τις εργασίες αύριο το πρωί στις 9 στην ίδια αίθουσα και κλεισμένων των θυρών με μια συνεδρίαση των συντονιστών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πάλι και κλεισμένων των θυρών ένα feedback ε, για τη δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου για την αναπτυξιακή συνεργασία και το απόγευμα στις, μάλλον όχι, στις 10 και 20 θα συνεδριάσουμε κανονικά και θα έχουμε έναν ε, μια συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 και την ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Καλό βράδυ και αύριο.